Colleghi, per favore, Καλό συνάδελφοι, για καθίστε. Πρέπει να αρχίσουμε έγκαιρα και να συνεχίσουμε επίσης έγκαιρα. Θα παρακαλέσω τους φωτογράφους και δημοσιογράφους να μην ε, καταλαμβάνουν θέσεις και να διευκολύνουν την αρχή των εργασιών μας να καλωσορίσω την κυρία Άστον, η οποία ελπίζουμε ότι θα μας βοηθήσει έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάντηση αυτή όχι μόνο για να γνωριστούμε περαιτέρω, αλλά για να παρουσιάσει τις κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της δράσης και επίσης για να έχει μαζί μας, και αυτή είναι μια δεύτερη ευκαιρία, μια ανταλλαγή απόψεων, τρίωρη ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι ε, μια σημαντική συμβή, στιγμή, συγγνώμη, μια στιγμή θα έλεγα συμβολική αλλά και υποδειγματική της ε, προσοχής την οποία έχει στρέψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις ακροάσεις αυτές. Η ίδια η κυρία Άστον αντιπροσωπεύει την καινοτομία πλέον της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης μέσω της εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας και μέσω του ρόλου που αναλαμβάνει όχι μόνο ως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και ως υπάτου εκπροσώπου της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Αντιπροσωπεύει πράγματι ένα στοιχείο καινοτομίας. Πριν να της δώσω το λόγο, να υπενθυμίσω στους συναδέλφους τους κανόνες της ακροάσεως αυτής. Θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί ε, γιατί ε, πρέπει να είμαστε αυστηροί για λόγους ανάγκης και όχι γιατί αρέσει στον Πρόεδρό σας. Ε, θα πρέπει να κλείσουμε τις εργασίες μας στις 4 το απόγευμα. Θα υπάρξει ένας πρώτος γύρος συζητήσεων όπου θα πάρουν τον λόγο οι συντονιστές της Επιτροπής. Θα υπάρξει επίσης η δυνατότητα να ακούσουμε και την αρχική απάντηση της υποψηφίας και θα ακολουθηθεί μια δευτερολογία. Θα ακολουθήσει μάλλον μια δευτερολογία. Επαναλαμβάνω ότι θα εφαρμόσω τους κανόνες αυστηρά. Θα έχετε και απευθύνομαι στα μέλη ένα λεπτό στη διάθεσή σας για να θέσει ο καθένας μία και μόνη ερώτηση. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο για να αποφύγω να σας διακόπτω. Η κυρία Άστον έχει πολύ λίγο χρόνο για να απαντήσει και θα πρέπει λοιπόν να περιοριστεί ο κάθε βουλευτή σε μία ερώτηση και αυτή η ερώτηση να διατυπωθεί παρακαλώ με ευκρινή τρόπο. Σας ευχαριστώ για το πνεύμα συνεργασίας που θα χαρακτηρίζει τις εντατικές εργασίες μας από εδώ και πέρα και δίδω αμέσως το λόγο στην κυρία Άστον για μια παρουσίαση η οποία δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τα 10 λεπτά. President. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι ενθουσιασμένη που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα για να συζητήσουμε τις προθέσεις μου ως πρώτη διπλοθεσίτησα της Ένωσης, δηλαδή υπάτη εκπρόσωπο εξωτερικών και πολιτικής ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ξέρετε εκτιμώ ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο. Η στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι ένα από τα κλειδιά των νέων μου ευθυνών. Η συνθήκη της Λισαβόνας έχει τεθεί πλέον ενισχύ και αυτό μας δίνει τεράστιες δυνατότητες. Υπόσχεται πολλά για το μέλλον των πολιτών της Ευρώπης και όλων όσων είχαν ζητήσει τέτοιες εξελίξεις από το Κοινοβούλιο. Μια πιο δημοκρατική ένωση και πιο αποτελεσματική στην οικονομία της και πάνω απ' όλα πιο αξιόπιστο ρόλο στον κόσμο. Συμβαίνουν μεγάλες αλλαγές αυτή τη στιγμή, σημειώνονται και κρίσεις και πρέπει η απάντησή μας να είναι ανάλογη. Λέω εμείς διότι είναι συλλογική η ευθύνη αυτή. Όπως πολλοί και από εσά είμαι πεπισμένοι ότι χρειάζεται και μέσα στην Ένωση και στον κόσμο περισσότερη δράση της Ευρώπης για την προώθηση της ειρήνης, την καταπολέμηση της ανέχειας και την απάντηση σε πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτή την πρόκληση πρέπει να την εξετάσουμε, να συνδυάσουμε την εταιρική σχέση με ηγετικό ρόλο, να προωθήσουμε τις αξίες μας και τα συμφέροντά μας, να ακούσουμε τι λένε οι εταίροι, μας, και όταν μιλάμε να ακούγεται η φωνή μας. Αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω, με τη βοήθεια όλων εσάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργαζόμενοι με τον πρόεδρο Μπαρόσο και άλλους συναδέλφους στην Επιτροπή ως ομάδα, και φυσικά και σε συνεργασία με την Προεδρία του Συμβουλίου. Ξέρω ότι ο νέος μου ρόλος σημαίνει τεράστιες ευθύνες και όλοι γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποτέλεσμα αυτόματα ή απλώς από την δήλωση προθέσεων. Θα κριθούμε από τα έργα μας. Πρέπει λοιπόν, οφείλουμε στους πολίτες μας και όλους όσους τρέφουν το βλέμμα τους προς εμάς να ανταποκριθούμε στις ευκαιρίες που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας Μία από τις μεγαλύτερες είναι η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Και αυτή θα είναι από τις υψηλότερες προτεραιότητες μου, θα σε εξηγήσω γιατί. Δεν είναι μία γραφειοκρατική δραστηριότητα άσκηση, αλλά μία μοναδική ευκαιρία να συνδυάσουμε όλες μας τις υποσχέσεις πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές για να εφαρμόσουμε μία συνεπή και ολοκληρωμένη στρατηγική. Πρέπει να δημιουργηθεί κάτι που να προσθέτει, να προσφέρει απτά στον πολίτη και να δείχνει στους μη Ευρωπαίους ότι είμαστε αξιόπιστος εταίρος. Από την Επιτροπή, το Συμβούλιο, τη Γραμματεία του Συμβουλίου πρέπει όλοι μαζί να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Έχει ήδη αρχίσει η δουλειά και εγώ ετοιμάζομαι για να Υποβάλλω πρόταση που να εγκριθεί από το Συμβούλιο τον Απρίλιο. Σε όλα αυτά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζωτικό ρόλο. Ήδη έχετε κάνει ορισμένες συμβολές και προσβλέπω σε στενή συνεργασία μαζί σας καθ' όλη αυτή τη διαδικασία. Όσο δημιουργείται όμως η υπηρεσία αυτή ακόμη, πρέπει εντωμεταξύ να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που τίθενται ήδη. Πρέπει να είμαστε ενεργοί για τα θέματα που αναμένουμε να κρίνει η Ευρώπη ή να κρίνουν την Ευρώπη. Ως πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες που έχουν εκφραστεί. Στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, το Ιράν, τη Μέση Ανατολή, τη Σομαλία και την Ιεμένη φαίνεται ότι υπάρχουν προτεραιότητες και προβλήματα. Έχω ήδη συμμετάσχει στην υπουργική διάσκεψη του ΝΑΤΟ για το Αφγανιστάν που μου έδωσε την ευκαιρία να συναντήσω τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Άντερς Ράσμουσεν και συμφωνήσαμε να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας πραγματιστικά για να υπάρξει μια πραγματική συνεργασία Ένωσης ΝΑΤΟ. Σκοπεύω να πάω στην Ουάσιγκτον σύντομα για να συζητήσω με την Χίλαρη Κλίντον για να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τις προσπάθειές μας για αυτά τα σφαιρικά προβλήματα και θα επισκεφθώ και τη Μόσχα και το Πεκίνο για τη Μέση Ανατολή θα συναντηθώ αύριο με τον γερουσιαστή Μίτσελ και τον Αντώνιο Μπλερ. Για το Ιράν οι υπηρεσίες μου είναι σε στενές επαφές με όλους τους παράγοντες που ενδιαφέρουν, που δρούν εκεί και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να απασχοληθούμε το θέμα της άρνησης του Ιράν να ανταποκριθεί στις διεθνείς του υποχρεώσεις. Εμείς στην Ένωση έχουμε μεγάλη ευθύνη για τις γειτονικέ μας χώρες. Αυτό είναι φανερό. Αλλά η διεθνής μας αξιοπιστία εξαρτάται και από τις σχέσεις αυτές καλής γειτονίας, δηλαδή πραγματικές πολιτικές μεταρρυθμίσεις στα Δυτικά Βαλκάνια έτσι ώστε όλη αυτή η περιοχή να μπορέσει κάποτε να ενταχθεί στην Ένωση. Έχουμε κάνει βήματα για να απελευθερωθούν οι θεωρήσεις με τη Σερβία, το Μοντενέγκρο και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Θα χρειάζεται και μια πραγματική στρατηγική για να αλλάξουν τα πράγματα στη Βοσνία ριζεγοβινη Πέρα από τα Βαλκάνια τώρα πρέπει να παίξουμε ενεργό ρόλο και στην Ουκρανία όπου προβλέπονται εκλογέ και θα υπάρξουν σημαντικά προβλήματα ιδίω για την ενέργεια. Η η Μολδόβα και οι χώρες του Νοτιού Καυκάσου επίσης ζητούν μεγαλύτερη δράση της Ένωσης. Γενικότερα η ευρύτερη μεσογειακή περιοχή επίσης είναι μεγάλη προτεραιότητα γιατί έχουμε ιστορικούς δεσμούς και κοινά συμφέροντα με τις χώρες της. Μεταξύ των προβλημάτων βέβαια είναι και η παράνομη μετανάστευση από τις χώρες αυτές. Και πέρα από την άμεση γειτονία μας στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική και στην Ασία για όλα αυτά πρέπει να επιδείξουμε καινοτόμο πνεύμα και αποφασιστικότητα. Εκτός από αυτά τα περιφερειακά θέματα έχω σκοπό να συνεργαστώ και για θέματα συγκεκριμένα όπως την μη διάδοση των πυρηνικών, την ε, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και κλιματολογικών αλλαγών. Αυτά δεν είναι μεμονωμένα θέματα, είναι τμήματα μεγαλύτερων, ευρύτερων προβλημάτων και πρέπει να λυθούν σφαιρικά. Το ίδιο και για τη διαχείριση των κρίσεων υπό την λεγόμενη κοινή πολιτική ασφαλείας και αμήνης. Ξέρω ότι σας ενδιαφέρουν πολύ και εσάς αυτά τα θέματα. Είναι θέματα που μπορούν να σώσουν ζωές, να ειρηνεύσουν περιφέρειες που αντιμετωπίζουν σειράξεις και είναι κάτι ζωτικό που μπορεί, στο οποίο μπορεί να συμβάλλει η Ευρώπη. Πρέπει βέβαια για όλα αυτά να έχουμε το κατάλληλο αριθμό προσωπικού και χρημάτων. Τέλος, κάτι για τις διεθνείς συμφωνίες. Τα πολύπλοκα προβλήματα ενός ενωμένου κόσμου απαιτούν πολύπλευρες απαντήσεις. Και για μένα αυτό ακριβώς σημαίνει βιώσιμη ασφάλεια. Για να το πετύχουμε χρειαζόμαστε εταιρικές σχέσεις με όλους τους παράγοντες, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία, αλλά επίσης Τουρκία, Ιαπωνία, Καναδά, Ινδία, Βραζιλία και Νότια Αφρική. Με τον ΟΗΕ, με τον ΝΑΤΟ, με την Αφρικανική Ένωση και πολλούς άλλους. Τέτοιου είδους σχέσεις η βελτίωση αυτών των σχέσεων θα είναι μεγάλο τμήμα της δραστηριότητάς μου ώστε να υπάρξουν οι κατάλληλες σχέσεις για να δοθούν κατάλληλες απαντήσεις στις προκλήσεις. Επίσης όμως πρέπει να καθοριστούν οι κανόνες με, την οποία θα, με οποίους θα εφαρμοστεί αυτή η διεθνή συνεργασία. Εδώ πρόκειται για μοναδική ευκαιρία. Μοναδική. Πρέπει να επιδείξουμε πνεύμα φιλόδοξο και τα λόγια μας να ακολουθούνται από πράξεις. Η συνθήκη του Λισαβόνας μας δίνει τις δυνατότητες αυτές. Και η δική μου δουλειά είναι να τα συνδυάσω όλα αυτά για να προμηθεύσω πνεύμα ηγετικό. Άρα χρειάζεται και η προσπάθεια η δική σας. Γι' αυτό θα είμαι υπόλογη για όλες μου τις δράσεις ενώπιόν σας και θα ζητήσω μεγάλες και ευρύτερες συζητήσεις μεταξύ όλων των παραγόντων της Ένωσης. Ευχαριστώ, αναμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Άστον. Θα περάσουμε τώρα στους συντονιστές. Υπενθυμίζω τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η συζήτηση σε μια πρώτη φάση. Ο μιλητής θα παρουσιάσει μία ερώτηση σε ένα λεπτό, θα ακολουθήσει η απάντηση της υποψηφίας για δύο λεπτά και θα υπάρξει ή ένα σχόλιο ή μια δεύτερη ερώτηση ενός λεπτού πάλιν. Και στο τέλος η κυρία Άστον έχει ένα λεπτό για να κλείσει την ερώτηση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μία ερώτηση ενός λεπτού. Ο κύριος Μπροκ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία υποψήφια, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που έχετε κάνει ενώπιον της Επιτροπής μας εξ ονόματος της ε, ομάδας του ΕΛΚ και φυσικά θέλω να εκφράσω και τις ευχές μου να μπορούμε να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία. Τώρα θα ήθελα να θέσω και ορισμένα ερωτήματα. Έχετε ένα δύσκολο καθήκον γιατί έχετε μεικτές αρμοδιότητες που εμπλέκουν και το Συμβούλιο και την Κομισιόν και είναι απαραίτητο να μπορέσετε να αρθρώσετε μια συνεκτική πολιτική που να εμπλέκει και τα δύο όργανα και αναφέρομαι ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Διπλωματική Υπηρεσία. Είσαστε διατεθειμένοι να δώσετε και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις απαραίτητες πληροφορίες και ενημέρωση για τα θέματα τα οποία άπτονται της ε, ε διπλωματικής υπηρεσίας. Θα αναλάβετε την πρωτοβουλία αυτή και δεύτερον βλέπετε το θέμα αυτό όπως και εμείς ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθούν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τον πολιετή σχεδιασμό. Τελείωσε ο χρόνος σας, ε, λέει ο Πρόεδρος. Αυτά ήταν τα ερωτήματα μου, λέει ο κ. Uh, σας ευχαριστώ για το πνεύμα αυτό, το επικοδομητικό μέσα στο οποίο και εγώ θέλω να κινηθώ και χαιρετίζω την δήλωσή σας. Εγώ πιστεύω ότι οι επικαλυπτόμενες αυτές αρμοδιότητες μπορούν να είναι κάτι θετικό και όχι κάτι το προβληματικό. Ακριβώς επειδή συνενούνται αυτές οι αρμοδιότητες, εγώ μπορώ να αναλάβω και τους δύο ρόλους με έναν τρόπο που θα εξασφαλίσει την εσωτερική του συνεκτικότητα έναντι του έξω κόσμου, αλλά και μέσα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αντιμετωπίζω λοιπόν το θέμα αυτό σαν μια πρόκληση προφανώς αλλά και σαν ένα πλέον έκτημα. Σε ό,τι αφορά τι αρμοδιότητέ μου και τι ευθύνε μου έναντι του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να παίξω και το ρόλο του Συμβουλίου και της Κομισιόν και εγώ θα είμαι ενώπιον του Κοινοβουλίου ως Επίτροπος, θα είμαι διαθέσιμη πάντα ενώπιον σας, αλλά θα σας δίνω και την προσθέμενη αξία του να εκπροσωπώ και το Συμβούλιο. Θα πρέπει να δούμε τώρα διαδικαστικά με ποιο τρόπο θα λειτουργήσει η επαφή μας. Γιατί ένα από τα θέματα τα οποία έχουν τονίσει ιδιαίτερα οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ότι είναι σημαντικές οι ευθύνε που έχει το αξίωμά μου και θα πρέπει να εξασφαλίσω ότι θα έχω τον απαραίτητο χρόνο για να έρχομαι ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν αυτά εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχή που θα έχω τη δυνατότητα να έρχομαι στο Κοινοβούλιο όσο το δυνατόν συχνότερα και να συνεργάζομαι μαζί σα για να αναπτύξουμε κοινέ δράσει και πολιτικέ. Ευχαριστώ. Ο Κυρία Άστον, δεν νομίζω ότι απήντησε στο θέμα των δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα του προπολογισμού και του ελέγχου του προπολογισμού σε ό,τι αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπου εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που έχουμε έναντι της Επιτροπής, άλλως αυτό θα σήμαινε μια υποβάθμιση των ελεκτικών δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύετε λοιπόν πρέπει να διατηρηθούν αυτά τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό και συμφωνείτε επίση ότι βάσει του άρθρου 22 η Κομισιόν θα πρέπει να έχει την αρμοδιότητα για τις εξωτερικές δράσεις πέραν της ΚΕΠΑ για όλες τις δράσεις που δεν έχουν να κάνουν με την ΚΕΠΑ και να υπάρχει η απαραίτητη παρουσία της ε, Κομισιόν σε όλα τα θέματα τα οποία άπτονται των εξωτερικών δράσεων, όπως παραδείγματος χάρη διαδικασία της Κοπενχάγης για το κλίμα. Αυτή είναι η ερμηνεία που έχετε εσείς σε σχέση με, το, με το ρόλο της Κομισιόν. Δύο υποδείγματα έχουν παρουσιαστεί. Αφενός υπάρχουν μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα θέλαν η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λειτουργεί μέσω της ε, Κομισιόν. Άλλοι θεωρούν ότι είναι ένα ιδιότυπο, ένα σουγγενές εγχείρημα και πρέπει να αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο. Σίγουρα ο προπολογισμό τη διπλωματική υπηρεσία θα υπόκειται σε απόλυτο κοινοβουλευτικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανεξάρτητα από τη διάρθρωσή του βάσει των δημοσιονομικών ε, κανόνων. Ο δικό μου ρόλο είναι να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει η σωστή ε, παροχή κονδυλίων ώστε αυτοί που χρειάζεται να πάρουν αυτούς τους πόρους είτε είναι πρέσβεις είτε είναι αντιπροσωπείς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν τη δυνατότητα μέσω αυτών των κονδυλίων να υποστηρίζουν τα σχέδια τα οποία θέλουμε να προωθήσουν. <clears throat> θα ήθελα τα χρήματα αυτά να να δοθούν στους πραγματικούς αποδέκτες προς όφελός τους και προς όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει φυσικά να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό. Αυτό είναι η πιο σαφής απάντηση που θα μπορούσα να σας δώσω. Ντίγκενινγκ, ένα λεπτό για μία ερώτηση, παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Άστον και θα ήθελα να καλωσορίσω από πλευράς των Δημοκρατών Σοσιαλιστών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να σας καλωσορίσω. Έχουμε ανάγκη από πολύ πιο αποτελεσματικές πολιτικές στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της ασφάλειας. Η συνθήκη της Λισαβόνα, έχει εισάγει κάποιες αλλαγές μεταξύ των οποίων και την δημιουργία της θέσης την οποία καλείστε να καταλάβετε. Συνδυάζεται λοιπόν, λέει ο κύριος Βιγγένη, τη θέση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με τη θέση του υπάτου εκπροσώπου για την εξωτερική πολιτική. Αυτό δεν θα πρέπει να είναι ένα τυχαίο, θα έλεγα, εγχείρημα, αλλά θα πρέπει να είναι μια συντονισμένη προσπάθεια βελτίωσης της ε, εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η δημιουργία επίσης ε, της νέας υπηρεσίας, της νέας εξωτερικής όπως λέγεται υπηρεσίας είναι μια προσπάθεια η οποία συνιστά κάτι το ιδιαίτερο καινοτομικό. Δεν, δεν διατυπώσατε κάποια ερώτηση. Αλλά παρόλα αυτά εγώ θα σεβαστώ τους κανόνες, λυπάμαι, δεν διατυπώσατε κάποια ερώτηση. Θέλετε κύριε Άστο να σχολιάσετε αυτά που είπε ο κύριος Βίγγενιν. It's... It's an additional challenge to try and guess the question. Πράγματι είναι, είναι μια επιπλέον προσπάθεια που πρέπει να κάνω να μαντέψω την ερώτηση. Παρ' όλα αυτά, δεν θα το κάνω αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω όμω κύριε Βίγκενινγκ εσεί προσπαθείτε να στρέψετε τη συζήτηση στι σχέσεις τις οποίε θα πρέπει να έχουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σχόλια γύρω από αυτό. Κάτι το οποίο έχω ήδη πει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αν θέλετε και την ανάπτυξη της δικής μου θέσης, του δικού μου ρόλου και της αντίστοιχης θέσης και ρόλου της εξωτερικής υπηρεσίας. Ε, πρέπει να διαβουλεύομαι με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν ληφθούν οι αποφάσεις από πλευράς του Συμβουλίου και θα πρέπει να είμαι όσο μπορώ παρούσα σε κάποιες συνεδριάσεις σας, ε, με τους περιορισμούς βέβαια, γιατί όπως ξέρετε θα έχω πάρα πολλή δουλειά. Βέβαια είναι αμφίδρομη η διαδικασία αυτή, ελπίζω να κατανοεί και να δέχεται το σώμα ότι θα πρέπει να μπορεί το Κοινοβούλιο και να μπορούν οι κοινοβουλευτικοί να συνεισφέρουν στην προβληματική των θεμάτων τα οποία θα με απασχολήσουν. Υπάρχουν και θέματα και ερωτήσεις όπως το πώς η εξωτερική υπηρεσία θα ε, στέκεται αρρωγός σε ε, βουλευτές που επισκέπτονται διάφορες περιοχές του κόσμου. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε και πώς ακριβώς θα υπάρχουν υπηρεσιακές επαφές ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη Νέα Εξωτερική Υπηρεσία. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία απαιτούν να υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει και να παίξει τον ρόλο τον οποίο καλείται να έχει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων Δεν ξέρω τώρα αν απάντησα στην ερώτησή σας αλλά κάποια προσπάθεια έκανα. Έχετε μία δευτερολογία κύριε Βίγκενινγκ ενός λεπτού. Είναι δύσκολο να μιλάει κανείς τη γλώσσα του από ό,τι φαίνεται λέει ο κύριος Βίγκενινγκ και θα συνεχίσω στην αγγλική. Περίπου τη μαντέψατε την ερώτηση η οποία ήταν πιο συγκεκριμένη. Ε, οι υψηλές θέσεις ε, ιεραρχικά εννοώ στην εξωτερική υπηρεσία θα πρέπει να περάσουν από ακρόαση ε, στις ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδιες όπως ή ε, εξωτερικών υποθέσεων, ανάπτυξης κτλ. Αυτό είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα διαβεβαιώσει για τις προθέσεις σας και τους Ευρωπαίους πολίτες η, συνέχεια στην ερώτηση, όχι η δεύτερη ερώτηση, η συνέχεια στην ερώτηση σχετικά με τις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να επικυρώνει τις συμφωνίες αυτές. Και μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν το διαβουλεύεται κανείς σχετικά με θέματα που αφορούν παράδειγμα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εδώ έρχεται η εταιρική συμφωνία με τη Λιβύη Κύριε Βίγενινγκ, ζήτω συγγνώμη για μια ακόμη φορά, αλλά ξεφύγατε χρονικά. Απάντηση ενός λεπτού από τη Βαρονιάστον. Θα σας απογοητεύσω σε σχέση με το πρώτο ερώτημα, γιατί δεν νομίζω ότι ο δρόμος αυτός τον οποίο αναφέρεται είναι ο καλύτερος σε ό,τι αφορά το προσωπικό και τη λειτουργία του. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι υψηλοί αξιωματούχοι, οι πεπειραμένοι αυτοί οι διπλωμάτες θα έχουν τη δυνατότητα να έρχονται και ενώπιον του Κοινοβουλίου. Ε, αυτή είναι η εντύπωση που έχω εγώ και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο. Σε σχέση τώρα με τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει των συνθήκων, αυτά τα θέματα τα έχουν εκφράσει πολύ πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα θέματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ακριβώς όπως προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Ναι, έτσι, για ένα λεπτό, μία ερώτηση και μόνο παρακαλώ. Κύριε Άστον, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μεταξύ των προκλήσεων που αντιμετωπίζετε, κύριε Άστον, φαίνεται ότι οι σημαντικότερε είναι καταρχήν να εξασφαλίσετε ότι θα διαδραματίσετε ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συντονίζετε τι δράσει των εμπλεκομένων για τα θέματα αυτά. Έχουμε τον πρόεδρο της Κομισιόν, έχουμε τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τους άλλους επιτρόπους οι οποίοι εμπλέκονται, κυρίως τον αρμόδιο επίτροπο για την πολιτική γειτονία και τη διεύνηση. Και η δεύτερη πρόκληση, όπως είπατε, είναι να μπορέσει να εκκινήσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, όπου θα χρειαστεί και εκεί να <clears throat> εξασφαλίσετε τον ηγετικό σας ρόλο έναντι των πολλών εμπλεκομένων και να έχετε μια σαφή σχέση μεταξύ του δικού σας γραφείου και του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας. Με ποιο τρόπο λοιπόν θα εδραιώσετε τον ηγετικό σας ρόλο σε αυτούς τους χώρους. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ίσως είναι λίγο ομό. Δύο λεπτά για να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ <clears throat> για το ερώτημά σας. Έχετε δίκιο όταν λέτε ότι υπάρχει μια πλειάδα ατόμων που έχουν διπλές αρμοδιότητες. Εγώ έχω εργαστεί για το θέμα αυτό τις προηγούμενες εβδομάδες πριν έλθω ενώπιόν σας και θέλω να σας τονίσω καταρχήν ότι η συνθήκη είναι απόλυτα σαφή σε σχέση με τις αρμοδιότητές μου. Η συνθήκη είναι εξάλλου το σημείο αναφοράς για όλους αυτούς οι οποίοι εξετάζουν το θέμα των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων. Οι συζητήσεις με τον πρόεδρο του, της Κομισιόν και του Συμβουλίου οδήγησαν σε μια σαφήνεια σε σχέση με τον εντοπισμό αυτών των αρμοδιοτήτων και αυτό είναι το δικό μου σημείο εκκίνησης. Δεύτερον, <clears throat> για να εξασφαλίσουμε μία συνεκτικότητα στο σύστημά μας, θα πρέπει να έχουμε μία δυνατότητα διαβούλευσης μεταξύ των θεσμικών οργάνων, ώστε να υπάρχει μία κοινή αντιμετώπιση. Αν δούμε λοιπόν το ρόλο των τριών επιτρόπων με τους οποίους εγώ θα συνεργαστώ πολύ στενά, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να εξασφαλίσουμε ότι είναι σαφείς οι αρμοδιότητες για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το στρατηγικό πλαίσιο, τη στρατηγική κατεύθυνση χάραξης πολιτικής με τη συμμετοχή του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. <clears throat> Ο στόχος είναι να μπορέσω σε συνεργασία με τους επιτρόπους να υλοποιήσω αυτές τις στρατηγικές κατευθύνσεις. Και έχω λοιπόν συζητήσει με τους τρεις υποψήφιους επιτρόπους και χωριστά και μαζί τους ως ομάδα και με τον πρόεδρο της Κομισιόν για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Έχουμε λοιπόν πολλά πρακτικά εγχειρήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρουμε. <clears throat> και σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, ο ρόλο μου είναι να προεδρεύω αυτού του Συμβουλίου και αυτό θα πράξω. Είναι πάρα πολλά τα οποία πρέπει να κάνω, αλλά υπάρχει σαφήνεια σε σχέση με το ρόλο. Ένα λεπτό δευτερολογία της κυρίας Νέιτς. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας, η οποία φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική. Να επανέλθω όμως σε αυτά τα οποία είπε ο προηγούμενος ομιλητές. Εξεπλάγην λίγο από την έλλειψη ενθουσιασμού την οποία επιδείξατε σχετικά με την δυνατότητα ακρόασης των υποψηφίων για τις ανώτερες θέσεις της εξωτερικής υπηρεσίας. Γιατί ο δισταγμός αυτός, από πού πηγάζει αυτός ο δισταγμός. Βεβαίως να το κάνω. Ε, δεν θέλω να απογοητεύω το κοινοβούλιο και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά κάποιες φορές φαίνεται ότι πρέπει να το κάνω. Η δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας είναι πράγματι κάτι το πολύ δύσκολο. Φυσικά έχουμε κόσμο εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο οποίος εργάζεται στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά επανειλημμένα και από ό,τι φαίνεται αυτές οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν επισκεφθεί πολλές φορές και το Κοινοβούλιο έχουν ικανοποιήσει τις περισσότερες φορές. Δεν θα ήθελα επίσης η διαδικασία επιλογής για τις ανώτατες θέσεις να είναι μια πολύ μακρόχρονη διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δημιουργήσουμε και να στήσουμε αν θέλετε το ταχύτερο δυνατόν και απαιτείται μια στρατηγική η οποία να είναι διαφανής, συνεκτική, να λαμβάνει υπόψη ε, τις ίσες ευκαιρίες ανδρών γυναικών κτλ. Μπραντνερ, ένα λεπτό μία ερώτηση. Καλώς ήλθατε, εξ ονόματος των Πρασίνων θα ήθελα να σας καλωσορίσω, κυρία Άστον. Έχετε ήδη αναφερθεί στο θέμα της ε, Λισαβόνας, της συνθήκης Λισαβόνας ότι γίνεται μια προσπάθεια να ξεπεραστεί η διφωνία Κομισιών και Συμβουλίου και εξάλλου για αυτό το λόγο υπάρχει το διπλό σας κασκέτο. Ένα σημαντικό τομέα τώρα σε όλα αυτά είναι τα θέματα της πολιτικής ε, γειτονίας. Θέματα όπως της Ουκρανίας, θέματα όπως ε, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το θέμα είναι πώς θα εξελιχθούν οι σημαντικές δράσεις που χρειάζονται και γι' αυτό είναι το ερώτημά μου. Για την, ε, για την πολιτική γειτονίας θα την διαχωρίσετε από τη διπλωματική υπηρεσία ή θα την αντιμετωπίσετε μαζί, η κυρία Αντιπρόεδρος, η κυρία Υποψήφια Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα σας εκπλήξει αυτό που θα σας πω ως απάντηση. Έχω συνεργαστεί με τον πρόεδρο της Επιτροπής για την υποβολή των προτάσεων του. Τη συζήτησε μαζί μου πριν τις εφαρμόσει. Αν εξετάσετε το ρόλο μου θα διαπιστώσετε ότι είναι σημαντικός, καλύπτει πάρα πολλά θέματα και ιδιαίτερα πρέπει να αποσαφηνίσουμε μερικά από αυτά, δηλαδή πώς θα εφαρμόσουμε τα προγράμματα που εγκρίνουμε. Μεταξύ των επιτρόπων λοιπόν με τους οποίους συνεργάζομαι θα καθορίσω συγκεκριμένες δικαιοδοσίες, θα έχουν και αυτοί οι ακροάσεις μαζί σας, θα τους ακούσετε, αλλά ο σκοπός μας είναι πρώτον για την ανάπτυξη να καταλάβουμε ότι είναι σημαντικό κάποιος να προσέχει την εφαρμογή των εκτελέσεων των ε, κονδυλίων του αναπτυξιακού αμύου, του ΕΤΑ. Για την πολιτική της γειτονίας εγώ έχω ταυτίσει τα προβλήματα και έχω πει ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει και εδώ να αποτελέσουμε πρωτοπορία. Η Επιτροπή δηλαδή με, αν με υποστηρίξει θα καταλήξουμε να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει με τις σχέσεις καλής γειτονίας και τρίτον θα υπάρχει κάποιος που θα ασχολείται με τον συντονισμό περιφερειακών οντοτήτων όπως ΑΣΕΑΝ και άλλων για να είμαστε βέβαιοι ότι ξέρουμε τι συμβαίνει και με τους οργανισμούς εκείνους. Αυτά. Ένα λεπτό για να απαντήσει η κυρία Μπραντνε. Εκπλήσω λιγάκι που λέτε ότι μπορείτε να αναλάβετε και θέματα της ε, πολιτικής γειτονίας. Εγώ δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρη αν αυτό είναι το θέμα, το, αν αυτές είναι οι αρμοδιότητες οι οποίες προκύπτουν από τη συνθήκη. Αλλά για την εξωτερική υπηρεσία το ερώτημά μου είναι θα συνενώσετε τις ενέργειες της ε, Κομισιόν με τις δράσεις της εξωτερικής υπηρεσίας. Και θα εξασφαλίσετε ότι θα λειτουργούν αρμονικά και σε συνεργασία οι αποστολές αυτές της ε, εξωτερικής πολιτικής και οι αποστολές των κρατών μέλων. Τι θα κάνετε λοιπόν εάν δεν υπάρξει η απαραίτητη συνεργασία στην περίπτωση αυτή. Έχετε την δυνατότητα να απαντήσετε για ένα λεπτό. Για το πρώτο ερώτημά σας. Εγώ δεν νομίζω ότι διαφωνούμε είναι πάρα πολλά τα οποία έχουμε να κάνουμε και εγώ δεν θέλω να επιλέξω μονάχα ορισμένου τομεί. Θα σα εξέπλητα αν ερχόμουν και δεν σα έλεγα ποιε είναι οι προτεραιότητέ μου, ιδίως στις αρχικές αυτές φάσεις του, του εγχείρηματος για την εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Εγώ θέλω να προωθήσω την πολιτική γειτονία μέσα στις δικές μου αρμοδιότητε, αλλά όπως ξέρετε υπάρχει και ένας επίτροπος ο οποίος θα αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Έχω έλθει σε επαφή μαζί του, είχαμε έντονε συζητήσει σε σχέση με το τι θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε, ιδίω σε ορισμένε περιοχές όπω αυτή της Βοσνίας, όπου πραγματικά εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για την τελμάτωση της πολιτικής κατάστασης. Νομίζω ότι η συνεργασία μας είναι θετική, είναι πλεονέκτημα και όχι μειονέκτημα και φυσικά ε, βασίζομαι στο γεγονός ότι το Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί πάντα τη δράση μας και θα εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα της. Ο κύριος Τάνοκ, Βαρονέσα Άστον λέει ο κύριος Τάνοκ, ήσασταν ταμείας ενός φορέα στη δεκαετία του 1970. Δεν έχετε ακόμα αποκηρύξει τις ε, δράσεις σας εκείνη την εποχή. Τώρα εσείς είστε αρμόδια για θέματα που είναι ακριβώς αντίθετα από την πολιτική αυτή για τον αφοπλισμό, θέματα δηλαδή εξωτερικής πολιτικής σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει δύο πυρηνικές δυνάμεις, την Αγγλία και τη Γαλλία και που είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα αγώνα εναντίον του ορολογίου στην περίπτωση του Ιράν που αναπτύσσει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υποστηρίζεται τη μονομερή, ε, το μονομερή πυρηνικό αφοπλισμό και σε σχέση με την ΚΕΠΑ πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα κοινό κέντρο επιχειρήσεων που να εδράζεται στις Βρυξέλλες για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν ήμουν πραγματικά τόσο ιδεαλιστική όσο με παρουσιάζετε. Η πραγματικότητα της δεκαετίας του 70, 1970 δεν είναι η πραγματικότητα της δεκαετίας του 2010. Οι προτάσεις τότε που είχαν τεθεί για αφοπλισμό ήταν σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο. Μπορείτε να προσπαθήσετε να απομονώσετε αυτό το στοιχείο. Εγώ ποτέ δεν υποστήριξα την εκστρατεία για, την, για τον ποινικό αφοπλισμό τα τελευταία 28 ή 30 χρόνια. Το δεύτερο ερώτημα που θέτεται που είναι πιο ουσιαστικό είναι το πώς θα αναπτύξουμε τις σχέσεις μας. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στο ΝΑΤΟ. Είναι πολύ σημαντικές σχέσεις με το ΝΑΤΟ και εγώ τόνισα στις αρχικέ μου παρατηρήσει, ότι μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για να μπορέσουμε να δούμε πώ μπορούμε να αναπτύξουμε μια πραγματιστική και δυναμική σχέση για το μέλλον. Κάτι το οποίο θα έχει μεγάλη σημασία για όλους μας. Σε ό,τι αφορά το να υπάρχει μια ενιαία δομή διοίκησης, εγώ δεν είμαι ακόμα πεπισμένη για την αναγκαιότητα μιας τέτοιας ε, δομής. Βάσει των συμφωνιών Βερολίνου ΣΥΝ, η συνεργασία μας με το ΝΑΤΟ, η δυνατότητά μας να λειτουργούμε με το ΝΑΤΟ και να χρησιμοποιούμε τους πόρους του ΝΑΤΟ φαίνεται ότι προχωρά πολύ θετικά και νομίζω ότι στις δύο περιπτώσεις που χρειάστηκε να κάνουμε κάτι τέτοιο ήταν θετικά τα αποτελέσματα. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι ακόμα βρισκόμαστε σε ένα σημείο που να απαιτείται νέα δομή. Μπορεί να υπάρχουν αποκλίνουσες απόψε κάτι μέλη και στο Κοινοβούλιο, αλλά εγώ θα ήθελα να σας πω ότι ακόμα δεν είμαι πεπισμένη για την ανάγκη μιας ενιαίας δομής για τα στρατιωτικά θέματα. Ο κύριος Στάνοκ έχει ένα λεπτό να θέσει συμπληρωματικό ερώτημα χωρίς μικρόφωνο, κύριο Στάνοκ. Χωρίς μικρόφωνο κύριε Στάρικ. Δεν μου δώσατε μια απάντηση ναι ή όχι για το αν υποστηρίζετε την, τον μονομερή πυρηνικό αφοπλισμό. Θα ήθελα μια απάντηση. Το επόμενο ερώτημα. Η Ινδία είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο και σημαντικό εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να ενισχυθούν περαιτέρω οι σχέσεις Ευρωπαϊκής ενωση Ινδία, ιδίως για τον αγώνα κατά του παγκόσμιου, της παγκόσμιας τρομοκρατίας που προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν που είναι γείτονε της ε, Ινδίας Πώ θα εξασφαλίσετε λοιπόν μια μεγαλύτερη συνεργασία στα θέματα αυτά και επίση θα ήθελα να ξέρω την προσωπική σα άποψη για το αν η Ινδία θα πρέπει να είναι μόνιμο μέλο του Συμβουλίου Ασφαλεία των Ηνωμένων Εθνών και αν ναι, ποιε άλλε χώρε θα πρέπει να είναι και αυτέ μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία κατά την άποψή σα και επίση για να συνεχίσω σε αυτό το πλαίσιο. Η κυρία Άστον για να. Πρέπει να απαντήσει η κυρία Άστον. Δεν είχε συμπληρωθεί το λεπτό. Μία ερώτηση, όχι περισσότερες ε, των, της μίας ερωτήσεως ε, στο λεπτό σας. Ε, θα μαντέψω το τέλος της ερώτησής σας. <clears throat> Νομίζω όμως ότι έπιασα, αν θέλετε, την ουσία. Νομίζω ότι η πολιτική της δεκαετίας του 70 δεν έχει νόημα σήμερα και δεν νομίζω ότι χρειάζονται να γίνουν πολλές συζητήσεις το ότι ήμουν ενθουσιώδης εναντίον της διάδοσης των πυρηνικών όπλων είναι κάτι που έχει σχέση και με τη σημερινή μου στάση για τον έλεγχο της διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι ανησυχούμε και εμείς και εσείς έτσι ώστε να ελέγξουμε τη διάδοση των όπλων αυτών μην διαπιστώστε φυσικά αυτά τα οποία ήμουνα στη δεκαετία του 70, αλλά μην κάνετε περισσότερες συζητήσεις χωρίς νόημα. Για την Ινδία, πράγματι η Ινδία παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό που έχει σημασία είναι πώς θα συνεργαστούμε επικοδομητικά με την μεγάλη αυτή χώρα. Συνάντησα τον πρόεδρο της ε, Ινδικής Ομοσπονδίας ε, επανειλημμένα, δεν είχα όμως τη δυνατότητα να συζητήσω τέτοιου είδους λεπτομέρειες για πιθανή συμμετοχή στο Συμβουλίο Ασφαλείας κτλ. Θα επισκεφθώ όμως την Ινδία το ταχύτερο δυνατόν. Ζητώ συγγνώμη, λέει. Στην κυρία Άστον, ο πρόεδρος, οι κανόνες ισχύουν και για σας. Ο κύριος Μελανσόν, ένα λεπτό στην εισαγωγή σας δεν αναφερθήκατε στην εταιρική σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε, η οποία έχει χαρακτηριστεί σαν κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό τον χαρακτηρισμό τον έχει δώσει και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν αναφερθήκατε επίσης και στη διαμόρφωση της μεγάλης διατλαντικής αγοράς τι θέση θα πάρετε στην εξέλιξη αυτής της πρωτοβουλίας και θα ήθελα να σας πω ότι εγώ προσωπικά βέβαια οφείλω να σας πω είμαι εναντίον αυτής της ιδέας. Δύο λεπτά η απάντηση της Αντιπροέδρου Άστον. Συστήνω τους συναδέλφους να στέκονται, να σέβονται μάλλον την ρύθμιση στην οποία έχω επανειλημμένα αναφερθεί. Διατλαντική αγορά, τι ακριβώς εννοείται να σας μιλήσω καταρχάς για τις σχέσεις με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Και ίσως να μην έχω απαντήσει πλήρως την ερώτησή σας, μπορείτε να επανέλθετε. Οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένε Πολιτείες είναι κρίσιμες σχέσεις. Είναι στρατηγική μας εταίρη σε αυτόν τον κόσμο. Πάντα είμαστε πλάι τους, σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου όπου απαιτείται να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος. Έχουμε διαφορετικούς ρόλους και διαφορετικές ευθύνες, παρόλα αυτά όμως η σχέση μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Ιδιαίτερα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε κάποιου συγκεκριμένου στόχου και μορφέ συνεργασία στρατηγικέ. Έχουμε το Συμβούλιο το Διατλαντικό, έχουμε το, ε, το Συμβούλιο Ενέργειας ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε, Έχουμε διαφορετικούς τρόπους και πλατφόρμες συζήτησης και όχι μόνο σε επίπεδο εμπορίου, αν και φυσικά ε, το ποσοστό του εμπορίου ανάμεσα στις Ηνωμένε Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστια σημασία και για αυτούς και για μας. Περιμένω την συγκεκριμένη ερώτηση. Κύριε Μελανσόν, δευτερολογία ενός λεπτού δεν γνωρίζετε τι είναι η διατλαντική αγορά. Να σας παραπέμψω σε, μία, σε ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παραπέμπει στη δημιουργία αυτής της αγοράς ήδη από το 2015. Σχετικά με το Αφγανιστάν, ξέρετε ότι είναι η πιο σημαντική ευρωπαϊκή στρατιωτική παρουσία από το δεύτερο πόλεμο και ε, πώς ακριβώς θα βοηθήσουμε για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε στο Αφγανιστάν, επαναλαμβάνοντας βέβαια ότι εγώ είμαι κατά της παρουσίας μας εκεί. Ένα λεπτό απάντηση της κυρίας Άστον. Σας ευχαριστώ να μου στείλετε το έγγραφο σχετικά με τη διατλαντική αγορά για το Αφγανιστάν. Ήμουν παρούσα όταν είχε παρουσιάσει ο αρμόδιος στρατιωτικός υπεύθυνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, τους στρατηγικούς στόχους στην χώρα αυτή. Το βασικό συστατικό είναι να προσπαθήσουμε να συνεισφέρουμε αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε καλύτερα και να υποστηρίξουμε μια αντίληψη βοήθειας του πληθυσμού και αυτό ακριβώς θέλει να προωθήσει και ο στρατηγός Κρίσταλ. Ήδη έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες τις οποίες μπορούμε να βελτιώσουμε. Η συνάντηση για το Αφγανιστάν στις 28 του μηνός στο Λονδίνο έχει πάρα μεγάλη σημασία για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Μπέλντερ, ένα λεπτό ερώτηση. κυρία υποψήφια αντιπρόεδρε της Κομισιόν, ως πρόεδρος αντιπροσωπείας θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με τον εβραϊκό χαρακτήρα του κράτους του Ισραήλ. Είστε αντιπρόεδρος της Κομισιόν, είστε και ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχετε αναφερθεί στον εγγενός εβραϊκό χαρακτήρα του Ισραηλού κράτους. Τι συμβαίνει όμως με την Παλαιστινιακή αρχή που ηγείται ενός αραβικού κράτους. Θα ζητήσετε από την Παλαιστινιακή Αρχή να αναγνωρίσει τον εγγενός εβραϊκό χαρακτήρα του κράτους του Ισραήλ. Γιατί αλλιώς θα υπάρξει σύγκρουση με τα ψηφίσματα του 1999 του ΟΗΕ. Η Άστον για δύο λεπτά. Αυτό το οποίο είμαι έτοιμη να πω είναι το εξής. Είναι κεφαλαιόδους χαρακτήρα να μπορέσουμε να έχουμε κάποια πρόοδο στη Μέση Ανατολή και να καταλήξουμε σε ένα καθεστώς δύο κρατών. Το κράτος του Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υφίσταται μέσα σε το πλαίσιο της ασφάλειας μέσα στην Μέση Ανατολή, όπως έχει και το Παλαιστινιακό κράτος. Πώς θα γίνει αυτό δεν θα το αποφασίσω εγώ. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί να εξετάζεται μεταξύ των δύο εμπλεκομένων και μέσα στη διεθνή κοινότητα. Προφανώς εγώ θα πρέπει να αντιμετωπίσω τα θέματα αυτά όταν επισκεφθώ τη Μέση Ανατολή που θα το πράξω όταν είναι κατάλληλες οι συνθήκες και όταν υπάρχει η δυνατότητα πρόοδου. Για μένα το πιο σημαντικό είναι όταν έχουμε αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες στο παρελθόν και περνάμε τώρα μια περίοδο νυνεμίας να μην θεωρούν οι πολίτες μας ότι αυτό είναι μια κατάσταση ασφάλειας και ηρεμίας. Αντίθετα, πρέπει αυτή η μικρή ανάπαυλα να μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε τη δυνατότητα ειρήνευσης ε, σας είπα ο κύριος Μίτσελ, ο κύριος Μπλερ θα είναι εδώ παρόντες ε, σύντομα εδώ στις Φρυξέλλες. Θα κάνουμε συναντήσεις στις λεγόμενες ομάδες του Παρισίου με στόχο να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες ελπίδες στην περιοχή αυτή και μια νέα όθηση για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ασφάλεια για όλους τους εμπλεκομένους. Κύριε Μπέλντερ, για ένα λεπτό. Το δεύτερο ερώτημά μου, κύριε Πρόεδρε, είναι το εξής δεν σας φαίνεται ότι είναι κατεπήγον να συγκαλέσετε μια διάσκεψη κορφής με το Ισραήλ το ταχύτερο δυνατό. Γιατί <clears throat> χρειάζεται να υπάρξει κατά την άποψή μου μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο για να ενισχυθούν οι αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ. Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι θέλει να διαδραματίσει ένα επιπροδευτικό ρόλο στη Μέση Ανατολή. Γι' αυτό δεν πιστεύετε κι εσείς ότι είναι επίγον να υπάρξει μια διάσκεψη κορφής για να υπάρξει σχέση εμπιστοσύνη με την νέα κυβέρνηση του Ισραήλ. Εγώ θα υποστήριζα λοιπόν κάτι τέτοιο, ώστε να μπορέσουμε με τον τρόπο αυτό να ενισχύσουμε τις σχέσεις οι οποίες ίσως δεν είναι ακριβώς στην καλύτερη κατάσταση.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 για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Άστον ανέφερε την κατάσταση που επικρατεί στο Ιράν και την θέληση της κυβέρνησής του να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια, πράγμα το οποίο είναι σημαντική απειλή και για το Ισραήλ και για τη Δύση. Μπορείτε να μας υποσχεθείτε ότι θα κάνετε ό,τι μπορείτε και όσο το δυνατόν συντομότερα, ό,τι είναι δυνατόν να γίνει, ώστε να αποφευχθεί αυτή η πιθανότητα. Το Ιράν δηλαδή να γίνει πυρηνική δύναμη. Είστε διατεθειμένοι, μπορείτε να μας το υποσχεθείτε εδώ και τώρα. Δύο λεπτά η πρόεδρο. I think it's, it's highly... Νομίζω ότι το Ιράν είναι προφανές ότι δεν δέχτηκε τη συμφωνία που του πρότεινε η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενεργείας και θα γνωρίζετε ότι πρόκειται για χώρα που έχει μεγάλη ιστορία, έχει κάνει λάθη αλλά αισθάνεται το ίδιο ότι έχει παρεξηγηθεί. Αν η χώρα αυτή θέλει να τύχει μεταχείρισης όπως αξίζει να έχει από την ιστορία της, τότε πρέπει να συνεργαστούμε μαζί της. Και εγώ καταδικάζω όλες τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυσικά είμαι διατεθειμένη για διάλογο. Αλλά δεν πρέπει να γίνει αυτό υπεκφυγή για να κερδιθεί χρόνος. Έχουμε επιδείξει πνεύμα υπομονής, κάναμε θετικές προτάσεις και ο κύριος Σολάνα έκανε προτάσεις. Είμαστε διατεθειμένοι λοιπόν για διάλογο αλλά με τις αρχές που θα μας είναι κοινά αποδεκτές. Και είμαστε, είναι σαφές το τι θέλουμε να είναι η εξέλιξη στο Ιράν. Και η διαδικασία 3 συν 3 θα μας δώσει προτάσεις και το Συμβούλιο θα αποφανθεί. Είμαστε λοιπόν σαφείς για το μέλλον που θέλουμε να έχει το Ιράν. Ένα λεπτό η απάντηση. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι κοινό και σαφής ο στόχο να μην γίνει πυρηνική δύναμη το Ιράν. Συμφωνούμε. Να μην έχει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αλλά αν ο Αχμαντίν Νετζάντ και επομένως και το Ιράν δεν σεβαστούν τις αποφάσεις των διεθνών οργανισμών. Είστε διατεθειμένοι να λάβετε σκληρά μέτρα κατά του Ιράν ως προς το Ισραήλ. Κυρία Αντιπρόεδρε. Το θέμα το οποίο θα συζητηθεί στα πλαίσια αυτής της δομής είναι θα έλεγα ο διτός τρόπος αντιμετώπισης του θέματος, τα πλαίσια στα οποία προανέφερα. Θα πρέπει να δούμε και τι άλλα μέτρα, οικονομικά κυρίως, θα ήσαν κατάλληλα για να ληφθούν. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεξάγουμε τις συζητήσεις μας και στο Συμβούλιο και στο μέλλον. Να πω επίσης, όπως είπα και στον κύριο Τάνοκ νωρίτερα, υπάρχει διάσκεψη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Τέλη της Άνοιξης, αρχές του καλοκαιριού. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία φε αυτής. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά για όλο τον κόσμο. Ας περάσουμε τώρα στη δεύτερη φάση. Πρόεδροι των υποεπιτροπών έχουν δικαίωμα παρέμβασης ενός λεπτού, θα απαντήσει για δύο λεπτά η υποψηφία και δεν θα υπάρξει δευτερολογία. Ξεκινάμε με την κυρία Άουταλα ένα λεπτό. Κυρία Άστον, μετά από την πρώτη συνάντησή μας και ανταλλαγή απόψεων έχετε επαναλάβει την πίστη σας στην λεγόμενη ήσυχη διακριτική διπλωματία για να ακουστεί η φωνή της Ένωσης στον κόσμο. Πώς θα γνωρίζουμε ότι αυτός δεν θα είναι ένας τρόπος για να μην θέτεται σημαντικά προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με χώρες στις οποίες έχουμε παράδοση σαν κοινοβούλιο να ξεκαθαρίζουμε τις απόψεις μας για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ιδιαίτερα στις χώρες στις οποίες διαπιστώνουμε σοβαρές παραβιάσεις θα ήσασταν διατεθειμένοι σαν παράδειγμα να συναντηθείτε με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες τις οποίες θα επισκεφθείτε που να εκπροσωπούν διαφορετικές φιλετικές ή εθνοτικές μειονότητες. Θα το κάνετε αυτό δημόσια, να σας πω και να απαντήσω άμεσα. Όταν μιλάω για την ήρεμη ε, διπλωματία, αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ θα είμαι ιδιαίτερα ήρεμη και ήσυχη πάντα. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι έχουμε την δυνατότητα, πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να συναντάμε τους ανθρώπους που μας ενδιαφέρουν χωρίς μεγάλη δημοσιότητα. Αυτό μπορεί να είναι ευεργετικό μερικές φορές. Και αυτό δίδει τη δυνατότητα σε πολιτικό επίπεδο για να καταλήξει κανείς τα απαιτούμενα συμπεράσματα. Μερικές φορές λοιπόν, και δεν σημαίνει ότι αυτό το έχουν κάνει οι προκάτοχοί μου, αλλά μερικές φορές το να φωνάζει κανείς και να γίνεται αντιληπτό στη διεθνή σκηνή, αυτό δεν βοηθάει πάντα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει στο τέλος να έχουμε πετύχει αυτό το οποίο επιθυμούμε να πετύχουμε και γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι στον κόσμο για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες για συγκεκριμένες χώρες. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να διαφοροποιήσω τις ε, μορφές παρέμβασής μου ανάλογα με τις χώρες. Κρίνοντας από το πόσο αποτελεσματικοί ήμασταν μέχρι τώρα και αν η στρατηγική την οποία ακολουθήσαμε ήταν σωστή. Σε καμία περίπτωση εγώ δεν εννοώ ότι θα αποκλίνω από την πεποίθησή μου για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που είναι ε, μια απόλυτη άποψη 100% αλλά σε επίπεδο μεθοδολογίας διαφοροποιούμε ίσως. Φυσικά και θα πρέπει να συζητήσουμε και με τις ΜΚΟ στην Ευρώπη για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάποιες από αυτές όπως η Λίμπερτη στο Ηνωμένο Βασίλειο τις γνωρίζω καλά. Υπάρχουν πολλές όμως στην Ευρώπη με τις οποίες θα ήθελα να συναντηθώ και να χρησιμοποιήσω την εμπειρογνωμοσύνη τους. Και φυσικά αυτό μπορεί να γίνεται και δημόσια όταν αυτό είναι χρήσιμο. Το λόγο έχει τώρα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας, ο κύριος Ντονζάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Άστον, θα επομιστείτε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, η οποία βασίζεται, πέραν των δράσεών της φυσικά, στις προσπάθειες που πρέπει να οδηγήσουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της. Μέχρι στιγμής είναι κάπως τα αποτελέσματα και αυτό αφορά τόσο και τα προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με ανάπτυξη βιομηχανικής ικανότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εσείς ως αντιπρόεδρος της Κομισιόν θα είσαστε οι αρμόδια και θα, φυσικά θα μπορείτε να δείτε όλα τα εγκάρσια διακυβευόμενα σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό, την εμπορική πολιτική, τη χρηματοδότηση για την αμυντική βιομηχανία μας και φυσικά και την έρευνα και την ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποιε είναι οι απόψεις για το θέμα αυτό. Έχετε το λόγο κύριε Αντιπρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Δύο σκέψεις καταρχήν. Ο Ευρωπαϊκός Φορέας Άμυνας και ο συντονιστικός του ρόλος. Το έχουμε δει αυτό ήδη στην περίπτωση των αποστολών που εμπλέκουν ελικόπτερα. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ περισσότερο και για την έρευνα και ανάπτυξη στα κράτη-μέλη και την ευκαιρία να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε προστιθέμενη αξία με το να έχουμε οικονομίες κλίμακος μεγαλύτερη συνεργασία των κρατών μελών. Ε, εγώ είμαι πεπισμένη με τις συζητήσεις που έχουν λάβει η χώρα μέχρι τώρα ότι αυτό είναι απαραίτητο. Από την πλευρά τώρα της Κομισιόν. Η Κομισιόν έχει την αρμοδιότητα για την έρευνα, την ανάπτυξη, την παιδεία, την κατάρτιση, όλα αυτά και όλα αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ευρύτερη προβληματική για το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε τις αμυντικές ικανότητες και πώς θα μπορούμε και πάλι να έχουμε μια στρατηγική σκέψη για το τι θέλουμε να κάνουμε στα θέατρα επιχειρήσεων. Θέλω λοιπόν να αναπτύξουμε περισσότερο τη σχέση μας με το ΝΑΤΟ και θα ήθελα να δω με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ πώς μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο αυτή η συνεργασία, φυσικά διατηρώντας τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν πώς θα έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία, πώς θα έχουμε καλύτερη ανάπτυξη σε έρευνα και ανάπτυξη, πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να ενισχύσουμε το ρόλο του αμυντικού φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τον κάνουμε αποτελεσματικό. Έχουμε... Έχουμε τελειώσει αυτή τη φάση με τους Προέδρους των Υποεπιτροπών. Περνάμε στη συνέχεια τώρα. Θα υπάρξουν παρεμβάσεις ε, ανά τρεις βουλευτές για ένα λεπτό ο καθένας, μία ερώτηση φυσικά στα πλαίσια του χρόνου που θα έχετε στη διάθεσή σας και για τρία λεπτά θα δώσει απάντηση στις τρεις ερωτήσεις η υποψηφία. Ξεκινάει ο κ. Σαλαφράγκα. Ο Μπόμπι Φίσερ, ο μεγάλος σκακιστής, κάποια στιγμή άδειασε την σκακέρα και είπε ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να ξεκινήσει μια νέα παρτίδα. Είναι σημαντικό λοιπόν το να μπορεί κανείς να προβλέπει τι θα κάνει ο αντίπαλός του και όχι μόνο ένα κακιστής αλλά και μια σημαντική πολιτικός όπως εσείς. Το ερώτημα είναι το εξή, κυρία Άστον. Πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να υπάρχει μια στρατηγική αντιμετώπιση ώστε η εξωτική μας στρατηγική να είναι συνεκτική με τις αξίες μας ορατή και αποτελεσματική για να ξεπεραστούν προβλήματα τα οποία είχαμε να δούμε αυτά που είδαμε χάρη το Δεκέμβριο όταν ορισμένα κράτη-μέλη δεν κράτησαν τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γενική Συνέλευση των Εθνών. και θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι ανάγκες σας σε επίπεδο προσωπικού και προπολογισμού για να επιτύχετε όλες αυτές τις, όλους αυτούς τους στόχους. Κύριε, κύριο Σάουιτ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ λέει ο κύριος Χάουιτ. Η... Οι συντηρητικοί κατηγόρησαν την κυρία Άστον και αυτό ουσιαστικά δείχνει που θέλουν να πάνε την Αγγλία εάν πάρουν ποτέ την εξουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βαρονέσα Άστον. Θέλω να χαιρετήσω αυτά που είπατε σε σχέση με τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των προτεραιοτήτων και ότι θέλετε να υποστηρίξετε απόλυτα αυτά που λένε οι συνθήκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όταν μιλάτε όμω για μια διαφοροποιημένη προσέγγιση στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία είναι οικουμενικά, πώ το εξασφαλίζετε αυτό, πώ εξασφαλίζετε ότι υπάρχει σαφήνεια στι ρήτρε των συνθήκων, αλλά διαφοροποιημένη εφαρμογή. Πώ θα βελτιώσετε την ασάφεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή πολλέ φορέ. Ο κ. Μποντή για ένα λεπτό κύριε Αντιπρόεδρε. Κατά την άποψή σας, ποιος είναι ο ρόλος τον οποίο θα πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ένωση για τη Μεσόγειο μέσα στα πλαίσια της αναζήτησης μιας λύσης για την κρίση της Μέσης Ανατολής. Αν δεν θέλουμε να, να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι μόνη οι οποίοι παρεμβαίνουν, οι Ηνωμένε Πολιτείε και ούτω ή άλλω δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχή, θα πρέπει η αλλω δεν ιδιαιτερα επιτυχη Ένωση να παίξει το ρόλο που τη αρμόζει στην Ισραηλο-Παλαιστινιακή κρίση. Ποιε είναι οι πρωτοβουλίε που προβλέπετε για να ευνοήσετε την δημιουργία ενό Παλαιστινιακού κράτου με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ω πρωτεύουσα. Τρία λεπτά για να απαντήσει η κυρία Αντιπρόεδρος, υποψήφια Αντιπρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ, <clears throat> κύριε Σαλαφράγκα. Είναι απαραίτητο να έχουμε μια ενιαία ενατένιση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αδειάσουμε προηγουμένως τη σκακέρα. Νομίζω ότι το έργο των προκατόχων μου ήταν εξαιρετικό. Έχουν επιτύχει πάρα πολλά και έχουν δημιουργήσει μια ισχυρή και θετική φήμη για, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα πρόσωπά τους σε όλο τον κόσμο. Πάντως, είναι απαραίτητο αυτή η εμπειρία να ενωθεί σε μία υπηρεσία και ένα άτομο, αλλά ένα άτομο το οποίο θα λειτουργεί ως κομμάτι μιας ομάδος. Πιστεύω ότι οποιοδήποτε ε, εκφράζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι ένα και το αυτό άτομο. Όχι 27 Υπουργοί, ο Πρόεδρος Κομισιόν, ο Πρόεδρος Συμβουλίου, οι βουλευτές δεν έχει νόημα. Χρειάζεται μία, μία φωνή για την Ευρώπη, η οποία να μιλάει με μία στρατηγική προσέγγιση. Αυτό είναι ο στόχο που θέλουμε να πετύχουμε. Σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό, εγώ είμαι ρεαλίστρια. Είμαι ρεαλίστρια σε σχέση με αυτά τα οποία θα δώσουν τα κράτη-μέλη στο μέλλον. Και στο βαθμό του δυνατό θα πρέπει να παραμείνω μέσα στα πλαίσια τα οποία έχουν προδιαγραφεί. Μπορούμε να επανέλθουμε αργότερα. Και για τον κύριο Χάουιτ. Ναι, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά, έχει τα απόλυτο δικαίωμα. Το μόνο που είπα είναι ότι η επίτευξη αυτού του επίπεδου οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων πολλέ φορέ απαιτεί διαφορετική προσέγγιση γιατί υπάρχουν διαφορετικοί πολιτισμοί και διαφορετικέ ιστορικέ εμπειρίε. Οι αντιπροσωπείε Ευρωπαϊκή Ένωση, οι υπηρεσίε εξωτερική δράση εδώ θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα κεφαλαιόδη ρόλο για να εξασφαλίσουν ότι θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τη στρατηγική μα σκέψη επιτοπίως και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να διασαφηνίσουμε τι ακριβώς θα πρέπει να κάνει η ενιαία υπηρεσία εξωτερικής δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να δώσει μια προσθέμενη αξία πέραν αυτού που κάνουν τα κράτη-μέλη. Η Ένωση για τη Μεσόγειο είναι ένα σημαντικό σώμα, αλλά έχει περάσει πολλές δυσκολίες γιατί δεν υπήρξε μεγάλη συμμετοχή από την αραβική πλευρά λόγω των προβλημάτων που γνωρίζουμε στην περιοχή της Παλαιστίνης. Υπάρχει η πρόταση για το κουαρτέτο, για να γίνει μια νέα, μια νέα συνάντηση του κουαρτέτου που προτείνεται από τη Ρωσία. Επομένως, <clears throat> ο συνδυασμός του ρόλου του κουαρτέτου και ο ισχυρότερος ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι το έναυσμα για μια περαιτέρω πρόοδο. Αλλά η Ένωση της Μεσόγειο αυτή τη στιγμή συνενώνει 40 κράτη της περιοχής που μπορούν να παίξουν ένα ρόλο. Νομίζω πρέπει να συνενώσουμε όλοι τις προσπάθειές μας για να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση στο Παλαιστινιακό πρόβλημα και νομίζω ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι ένα καλό σημείο κίνησης. Κυρία Ντεκάιζερ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Άστον, μας θυμήσατε σε ποιο βαθμό επιθυμείτε να ακολουθήσετε μια πολιτική στοχευμένη στο αποτέλεσμα. Και ήδη τον μήνα Δεκέμβριο μας είχατε υπενθυμίσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και μας είπατε ότι ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση και να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Επανέρχομαι λοιπόν στην ερώτηση Μποντής. Πώς θα το κάνετε αυτό σχετικά με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που αφορούν τη Λωρίδα της Γάζα, την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Πώς θα πετύχετε αποτελέσματα, θα συναντηθείτε με τον κύριο Μπλερ. Μα τον Μπλερ τον διόρισε ο Μπούς σε επίπεδο κουαρτέτου. Εσείς ελπίζω σαν γυναίκα και σοσιαλίστρια θα διοριστείτε από εμά. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Ο κύριος Μπλερ δεν πέτυχε τίποτα. Εμείς περιμένουμε αποτελέσματα από εσά και θα ήθελα να μάθω ποιους δρόμους θα ακολουθήσετε για να τους πετύχετε. Ο κύριος Σάουλ και ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Υποψηφία, σύμφωνα με το Κοινοβούλιο, η ενεργειακή σας πολιτική είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής. Και ερώτω, πώς προτίθεστε να πείσετε τη Ρωσία να μην χρησιμοποιήσει τα ενεργειακά της αποθέματα ως εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής έναντι άλλων χωρών. Και πώς θα προστατεύσετε τους ανατολικούς μας γείτονες από την κατά της υποβολής τέτοιων πολιτικών πιέσεων μέσω της ενεργείας. Νικολάη, ένα λεπιτό. Ευχαριστώ. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση και ελπίζω να λάβω συγκεκριμένη απάντηση. Αφορά το Αφγανιστάν. Βασίστηκα στη γραπτή σας απάντηση. Ποια νομίζετε ότι πρέπει να είναι η επόμενη φάση της ε, δράσης μας για το Αφγανιστάν. Ανταπάντηση. Ε, κοιτάξτε, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Κυρία Ντεκάιζερ, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει να υπάρξουν απτά αποτελέσματα και η απογοήτευση που αισθάνεστε και εσείς και άλλοι μπροστά στην έλλειψη αποτελεσμάτων σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι δικαιολογημένη. Το Συμβούλιο είπε ρητά ποιες είναι οι προθέσεις μας και επομένως για μένα αυτό που χρειάζεται είναι πώς θα πραγματοποιηθούν οι στόχοι αυτοί. Τι νομίζουμε ότι μπορούμε να κάνουμε αλλά και τα υπόλοιπα. Εγώ δεν θεωρώ ότι επειδή θα υπάρχει, θα είναι και αύριο ο κύριος Μπλερ παρόν θα μου λύσει εκείνος τα προβλήματα, εγώ θα τα λύσω. Και ήδη έχω αρχίσει να συζητώ με την Υπουργό Κλίντον, αλλά δεν πρόκειται να σας δώσω τώρα μια βιαστική λύση πριν γνωρίσω ακριβώς πού θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Αλλά πρέπει να είναι σαφές ότι όταν το αποφασίσω θα το πράξω και θα αναφέρω τακτικά στο Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Αφού μάθω, επαναλαμβάνω, ποια είναι ακριβώς τα προβλήματα και τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε. Έτσι ώστε τα χρήματα που θα βάλουμε στην περιοχή εκείνη να φέρνουν κάποιο απτό αποτέλεσμα. Κύριε Βόλσκι, μιλήσατε για εξωτερική πολιτική της Ρωσίας μέσω της ενέργειας. Καταρχήν, πρέπει να έχουμε μια στεναρή σχέση με τη Ρωσία αλλά και δική μας ενεργειακή στρατηγική που να μας επιτρέπει να διαφοροποιούμε τις πηγές μας ώστε να μην εξαρτόμαστε παραπάνω από τη Ρωσία γιατί η εξάρτησή μας είναι ήδη κατά 50% από αυτήν. Η διαφοροποίηση λοιπόν των πηγών μας και χρησιμοποίηση διαφορετικών πηγών ενεργείας ηλιακή, αιωλική και άλλες καθώς και η δημιουργία διαφόρων αγωγών. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι μερικά από αυτά τα θέματα είναι καθαρά πολιτικά και όχι οικονομικά και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε στη Ρωσία να πάψει να τα θεωρεί πολιτικά. Εντάξει για το Ουκρανία τα είπατε όλα αυτά θα επανέλθω. για το Αφγανιστάν ποιο πρέπει να είναι το επόμενο βήμα. πρέπει να τονίσουμε τις επιτυχίες που είχαμε σημειώσει, παραδείγματος χάρη στα υγειονομικά από το 2002. Αλλά υπάρχουν και άλλα προβλήματα βέβαια και θα ήθελα να υπάρξουν απτά αποτελέσματα για τον λαό του Αφουγανιστάν. Μάουρο για ένα λεπτό. Presidente, signora... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Άστον, σχετικά με την υπόθεση την οποία κυκλοφορούν ορισμένοι, ότι θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μία θέση από κοινού, μία έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ποιες είναι οι δυνατότητες τις οποίες έχετε ακούσει από τα κράτη-μέλη και θεωρείτε την πιο πιθανή και ποια στρατηγική θα ακολουθήσουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχουμε τον συγκεκριμένο στόχο. Κύριο Πεγιό, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Άστον. Έχετε επανέλθει ήδη στην Ένωση για τη Μεσόγειο και η Ισπανική Προεδρία θεωρεί ότι είναι μια βασική προτεραιότητά της. Όπως γνωρίζετε, τον μήνα Ιούνιο θα γίνει μια σημαντική συνάντηση όπου θα συζητηθεί η, εναλλακτική μορφή λειτουργίας και συνέχιση των δραστηριοτήτων της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Πώς θα ξεπεράσουμε ε, τις δυσκολίες που είχαμε μέχρι τώρα και πώς θα σεβαστείτε την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ευρωμεσογειακής χωρίς να αφήξουμε τις πιστώσεις της διαθέσιμες για την πολιτική γειτονίας. Σούλτς ένα λεπτό. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία για το σημαντικό και δύσκολο καθήκον σας και θεωρώ δεδομένο ότι παρά το γεγονός ότι δεν έχετε αρμοδιότητες ιδιαίτερες στην πολιτική γειτονία ότι σίγουρα θα αναλάβετε πλήρως την ευθύνη της πολιτικής για την Ρωσία. Έχει διαπιστωθεί ότι εκεί στην πολιτική γειτονία βρίσκονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς θα ακολουθήσετε την πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προχωρήσουμε προς μια εξυγχρονισμένη σχέση εταιρικού χαρακτήρα και μπορείτε να μας περιγράψετε τη νέα μορφή που θέλετε να έχει η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό και επίσης για τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τι ακριβώς θέλετε να διαγράψετε ως κατεύθυνση. Τρία λεπτά για να απαντήσει η υποψήφια κυρία Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Το ερώτημα μου πρώτο ερώτημα ήταν πολύ απλό. Δεν ξέρω. Για το λόγο γιατί αυτό το θέμα τις τελευταίες πέντε εβδομάδες που ασχολήθηκα με τα ζητήματα αυτά δεν πέρασε καν το μυαλό μου. Με πιάσατε λοιπόν να υπάρχει αυτό το θέμα κύριε Μάουρο για το οποίο εγώ δεν έχω καμία απάντηση. Δεν είναι ένα θέμα για το οποίο δεν πρέπει να σκεφτούμε. Αλλά υπάρχει τώρα μια πλειάδα διαφορετικών απόψεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ζήτημα αυτό. Αυτό που είναι αποτελεσματικό, που είναι απαραίτητο βέβαια, θα ήταν να μπορέσει να υπάρχει κάποια διαβούλευση στην, ε, στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτή τη βδομάδα. Θα είμαι ειλικρινή μαζί σα, δεν ξέρω ακόμα. Ένωση για τη Μεσόγειο. <clears throat> Όπως βλέπω αυτή τη στιγμή την κατάσταση αυτή, βέβαια αυτά είναι μια συνέχιση της διαδικασίας της Βαρκελόνης, που ήταν ε, ένα σύνολο από ενδιαφέρομενες χώρες της Μεσογείου, και το πιο ενδιαφέρον που προέκυψε ήταν η παροχή πόρων για διάφορα σχέδια περιφερειακού χαρακτήρα, ενέργεια, παιδεία κτλ. Θα πρέπει να περιμένουμε όμως να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το σύνολο των εγχειρημάτων. Με το τέλος της κοινή προεδρίας Αιγύπτου και Γαλλίας θα τεθούν ερωτήματα για τη συνέχεια. Και εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε και καλύτερα ποιος θα είναι ο ρόλος, αν υπάρχει κάποιος τέτοιος ρόλος, του προ, της Προεδρίας του Συμβουλίου. Αυτή η συζήτηση δεν έχει λάβει ακόμα χώρα. Αυτό το οποίο θέλω να εξασφαλίσω είναι ότι θα πρέπει να είναι πραγματικά αποτελεσματική η Ένωση για την Ευρώπη. Εάν υφίσταται θα πρέπει να είναι αποτελεσματική. Τα πράγματα φαίνεται να βελτιώνονται, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι συναρμόζεται με τη γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ένωση για τη Μεσόγειο. Είναι σημαντικό λοιπόν, ακόμα και αν είναι μια εταιρική σχέση, να έχει καλή συναρμογή με τις άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια. Για το ερώτημα του κύριου Σούλς. Έχουν πει πάρα πολύ ότι έχουμε μια μορφή επικάλυψης, αλλά εγώ το βλέπω σαν μια συνεργασία. Στις ε, λίγες αυτές περιπτώσεις που εγώ βρέθηκα σε συναντήσεις με κορυφής με τη Ρωσία, ιδιαίτερα με τον πρόεδρο Μέτβεντεφ, υπάρχει αυτή η συζήτηση για μια εταιρική σχέση για το μέλλον. Βρισκόμαστε τώρα στη φάση που προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε τη συμφωνία για την εταιρική σχέση. Δεν έχουμε προχωρήσει ιδιαίτερα σε ορισμένου τομεί αυτή τη ε, συμφωνία και όπω φαντάζεστε, τα ανθρώπινα, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τμήμα του έργου μας. Αλλά σας λέω και πάλι το σημαντικό είναι να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να θέτουμε αυτά τα ζητήματα και να θεσπίσουμε τους μηχανισμούς που θα μας οδηγήσουν σε αποτελέσματα. Αυτό είναι αυτό που με ενδιαφέρει, το τελικό αποτέλεσμα και πώ θα το επιτύχουμε. Θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να θέτουν μία ερώτηση στο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους για να υπάρχει και η κατάλληλη απάντηση. Ο κύριος Βανόρντεν για ένα λεπτό έχει το λόγο. Κύριε Άστον, όπως γνωρίζετε, είχα ευθύνε στα πλαίσια της διεξαγωγής των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Εσείς έχετε επισκεφτεί τέτοιου είδους επιχειρήσεις εκτός φυσικά από την περιοχή που σας ενδιαφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σχετικά με τις στρατιωτικές δυνάμεις που έχουμε στο Αφγανιστάν. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δυνάμεις φυσικά στο Αφγανιστάν. Θα πανά όμως πολλά χρήματα εκεί. Ξέρετε πόσα χρήματα δαπανώνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν κατέτος και τι βήματα ε, θα αναλάβετε έτσι ώστε τα χρήματα αυτά να μην πέφτουν, ε, να μην γίνονται αντικείμενο κατάχρησης. Κυρία Όμεν Ρόιτεν, ένα λεπτό. Είπα Όμεν Ρόιτεν. Κυρία Άστον, αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιόν. Εσείς τι θα κάνετε, προς ποιον θα είστε πιστότεροι. Δύο παραδείγματα για το Ιράκ. Τι φρονείτε για τον πόλεμο στο Ιράκ, δικαιολογείτε ή όχι. Και δεύτερον, η χάρτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δύο χώρες μέλη δεν την συνυπέγραψαν. Τι φρονείτε. Χάρτα ανθρωπίνων δικαιωμάτων λέγω. Πεντζέρι. Ευχαριστώ κύριε Άστον. Φανταζόμενος ότι η εξωτερική πολιτική και η πολιτική γειτονία ανήκουν σε μια ενωτική στρατηγική εξωτερική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται με τις σχέσεις μας με τις χώρες του Μαγκρέμπ. Έγινε ένα σημαντικό βήμα με την υιοθέτηση ενός κοινού ανακοινωθέντος για το Μαρόκο και καθορίζεται η οδός που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων και τη συμφωνία την εταιρική. Προβλέπεται επίσης και η δημιουργία μιας συνάντησης κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαρόκου. Τι μπορεί να προσφέρει η συζήτηση σε αυτό το στόχο και ο στόχος αυτός μπορεί να είναι χρήσιμος και για τις υπόλοιπες χώρες του Μαγκρέμπ. Έχει το λόγο η κυρία Άστον για να απαντήσει σε τρία λεπτά στις τρεις ερωτήσεις. Κύριε Βανόρντεν, νομίζω ότι αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε στο Αφγανιστάν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Είναι βασικό να καταλάβουμε γιατί είμαστε εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει τον ρόλο που καλείται να παίξει στη διαδικασία αυτή. Δεν έχω ακριβώς τις πιστώσεις για φέτος, αλλά έχω κοιτάξει το κόστος όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια και είπα ότι αφιερώνουμε πάρα πολλούς πόρους και έχουμε γενικά μια οικονομική στενότητα και αυτό καθιστά τις προσπάθειές μας σε άλλους τομείς πιο δύσκολες. Υπάρχουν πάντως ε, ενδείξεις οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχουν όλο και λιγότερες καταχρήσεις των κοινοτικών χρημάτων στη χώρα αυτή και τα, οι πιστώσεις οι κοινοτικές γίνονται όλο και πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε έστω και παρέχοντας τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία συνδέονται ε, με την βοήθειά μας στον τομέα της πολιτικής, στον τομέα τον κοινωνικό, το οικονομικό και όχι αυστηρά το στρατιωτικό. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία και έτσι θα συνεργαστούμε μεταξύ μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για την κυρία Όμεν Ρόιτερ. Το βασικό θέμα είναι να μην έλθω ποτέ σε αυτή τη θέση. Το θέμα είναι να προσπαθήσω να συνδυάσω το Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο με τη δική σας βοήθεια πάντα, έτσι ώστε να υπάρξει μια κοινή στρατηγική αντίληψη. Η εμπειρία μου μέχρι τώρα, όταν συμμετείχα για τρία χρόνια στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης, είναι ότι υπάρχει καλή θέληση έτσι ώστε να καταλήγουμε στα σωστά συμπεράσματα και μπορώ να το μαρτυρήσω αυτό και για το Συμβούλιο ε, Εξωτερικών Υποθέσεων. Πρέπει να ακολουθήσουμε και να επιδιώκουμε πάντα την κοινή πολιτική και πρέπει φυσικά να μην καταλήγουμε στον κατώτερο πάντα κοινό παρανομαστή αλλά στον υψηλότερο αν είναι δυνατόν για να πετύχουμε τους στόχους μας. Σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράκ. Εγώ όταν ξεκίνησε ο πόλεμος ήμουν ένα μέλος της κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με βάση αυτά που γνώριζα τότε ήμουν πεπισμένη ότι καλά κάναμε και ενεπλάκημεν. Ναι, Το τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα είναι να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα των δομών και της λειτουργίας της χώρας αυτής. Πρέπει να είμαστε στραμμένοι στο μέλλον, πρέπει να στηρίξουμε την σταθερότητα, την ευημερία, την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τομεί στους οποίους έχουμε ε, πεποίθηση ότι πρέπει να προωθήσουμε. Γκάλερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Βαρόνι Άστον. Εδώ και δέκα χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να έχω απάντηση στο ερώτημά μου. πέρασε ο καιρό. ο χρόνος ίσως θα μπορέσει να απαντήσει σε ένα άλλο πλαίσιο η κυρία Άστον. Θα βρούμε έναν τρόπο να σας δώσει μια απάντηση ίσως με άλλο τρόπο, αλλά εγώ πρέπει να διαχειρίζομαι με αυστηρότητα το χρόνο αυτό. Ναι, είναι σημαντικό και για τι χώρε του Μαγκρέπ, θα απαντήσει η κυρία Πίτροπος. Κύριε Γκάλερ, για ένα λεπτό. Εδώ και δέκα χρόνια έλεγα, κυρία Αστόν υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Από το 2003 έχουμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας η οποία έχει ενημερωθεί το 2008 και έχουν συγχωνευτεί οι φορείς ε, σχεδίασης. Παρ' όλα αυτά τα εθνικά κράτη-μέλη κάνουν τη δική τους πολιτική η οποία πολλές φορές υποσκάπτει την ε, στάση της, της, τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε την πρόθεση να προχωρήσετε σε μια λευκή βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Μήπως θεωρείτε επίση ότι είναι λογικό τα στρατιωτικά και πολιτικά σχέδια να εφαρμόζονται μέσα από ένα ευρωπαϊκό επιτελείο και όχι να περιμένουμε τα κράτη-μέλη να δώσουν τα δικά τους επιτελεία για την πρακτική εφαρμογή αυτών των σχεδίων. Κύριος Κάτσιν για ένα λεπτό. Στις αρχές Δεκεμβρίου καταθέσαμε μία ερώτηση σχετικά με τον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Αναφερθήκατε στα θέματα ασφαλείας τότε και σταθερότητας, η κατάσταση όμως έχει χειροτερεύσει από τότε και πρέπει να υπάρξει μια περαιτέρω παρέμβαση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε να πετύχουμε τον πολιτικό συμβιβασμό. Όλε οι προθεσμίε που είχαμε θέσει έχουν πλέον περάσει. Οδηγούμεθα στην ανεξαρτησία τη Ρεπούμπλικα Σέρβσκα. Μπορεί να γίνει δημοψήφισμα το οποίο θα έχει σαν συνέπεια τη διάλυση της Βοσνίας Ευζεγοβίνης, κάτι το οποίο θα προκαλέσει πάρα πολλά μεθοριακά προβλήματα. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν και σε μια φάση, σε ποια φάση μάλλον, στα πλαίσια της διαχείρισης της κρίσης στη Βοσνία. Θυμίζω ότι φέτος θα γιορτάσουμε δυστυχώς την 15η επέτειο της φαγής της Ρεμπρένια. Κύριο Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω και εγώ την αντίθεσή μου με την υποψηφιότητα της κυρίας Άστον γιατί ακριβώς εξυπηρετεί την πολιτική της Λισαβόνας για την οποία ε, εκφραστήκαμε αρνητικά πολλαπλώς. Η απάντηση της κυρίας Άστον όμως στο ερωτηματολόγιο του Κοινοβουλίου και μάλιστα στο σημείο 3 νομίζω μας δικαιώνει πλήρως. Θέλω να μου πει η κυρία Άστον γιατί δεν είναι διατεθειμένη να παρέχει στο Ευρωκοινοβούλιο πληροφορίες και έγγραφα σε ίση βάση με το Συμβούλιο. Σε αυτή την ερώτηση η κυρία Άστον δεν απάντησε. Και επίσης θα ήθελα να μου πει τι προτίθεται να κάνει ώστε να αλλάξει η απαράδεκτη κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Κούβα, ώστε να υπάρχουν ομαλές σχέσεις με αυτή τη χώρα και γενικά να σημειώσω, ευτυχώς λέω εγώ, η κυρία Άστον δεν τοποθετήθηκε καθόλου στο θέμα των σχέσεων με τη Λατινική Αμερική. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Τρία λεπτά η κυρία Άστον. Ξεκινώ με τον κύριο Παντσέρη, γιατί νομίζω ότι δεν του έδωσα πλήρη απάντηση και λυπάμαι. Ξέχασα από τις σημειώσει μου να πω το εξή. Για τη διάσκεψη με το Μαρόκο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο σχέδιο, αλλά σίγουρα πρέπει να έχουμε στενότερη επαφή με τις χώρες του Μαγκρέμπ και να σκεφτούμε το θέμα αυτό του Μαγκρέπ μέσα στην πολιτική <clears throat> γειτονία και επέκεινα. Για τον κύριο Γκάλερ. Για το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή για τη δυνατότητα να έχουμε μία λευκή βίβλο. Θα πάρω και περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Τώρα, για το να προχωρούν τα κράτη-μέλη σε ενέργειες μόνα τους. Τα κράτη-μέλη έχουν και αυτά αρμοδιότητες στον αμυντικό τομέα. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε όταν λέτε ότι κάνουν του κεφαλιού τους τα κράτη-μέλη πολλές φορές. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και να επιτύχουμε κοινά αποτελέσματα. Στα θέματα της διοίκησης Άμα πάρετε την περίπτωση του Northwood και τον ε, Ναύαρχο Χάτσον για τη Σομαλία, εκεί ήταν εποφελής ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι πόροι από τα κράτη-μέλη και χωρίς αυτό να ενσωματωθούν αυτοί οι πόροι σε μια ευρωπαϊκή δομή. Νομίζω λοιπόν ότι μέχρι στιγμής λειτουργεί αυτό το σύστημα. Για τη Βοσνία, κύριε Κέλλιν, έχετε απόλυτο δίκιο, υπάρχουν πραγματικά ζητήματα που πρέπει να τα αντιμετωπίζουν. Ο κ. Βαλστίνσκο και εγώ έχουμε συναντηθεί πολλές φορές και πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με άλλους για να σκεφτούμε ποια είναι η στρατηγική μας εκεί. Εδώ έχουμε μια χώρα με διαφορετικές εθνοτικές κοινότητες που θα πρέπει να συμβιούν διατηρώντας την εθνοτική τους υπερηφάνεια. Μπορούμε να κάνουμε όσα δημοψηφίσματα θέλουμε, αλλά πρέπει να δημιουργηθεί και ο ιστός μιας χώρας. Πώς θα γίνει αυτό όμως, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Οι εκλογές στη Βοσνία θα γίνουν τον Οκτώβριο. <clears throat> θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι όπως έλεγε ο Λόρδος Άσταουν ότι η προοπτική της ε, ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο συνδετικός ιστό που κρατούσε ενωμένη την Βοσνία και ο κ. Βαλεντινέσκο το επιβεβαίωσε. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουν όλοι στη Βοσνία τι μπορεί να του δώσει η Ευρώπη και ποια είναι τα ωφέλη που μπορούν να αποκομίσουν. Πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε μονάχα την επαφή με του πολιτικούς ηγέτες και να εξηγήσουμε και στο λαό της Βοσνίας τι μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να ζήσουν σε ειρήνη και να αποκομίσουν τα θετικά αποτελέσματα της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω είμαι σε επαφή με την Βοσνία και τον κύριο Βαλεντινέσκο και του δίνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη. Σε ό,τι αφορά τώρα τα ερωτήματα που θέσατε, που ήταν τέσσερα, για τη συνθήκη της Λισαβόνας, έχετε και εσείς αρμοδιότητές σας. Τώρα, για τα έγγραφα του Συμβουλίου, εγώ είμαι έτοιμη να σας δώσω πληροφορίες, αλλά υπάρχουν και κάποια όρια για το πότε μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες και πότε όχι για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ θα πρέπει να δούμε αν λειτουργεί αποτελεσματικά η στρατηγική μας για την Κούβα, αλλά είναι γεγονός ότι εξακολουθούν να παραμένουν πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα στη χώρα αυτή. Εάν σας τίθεται κυρία Άστον, τίθεται άνω της μία ερωτήσεις έχετε δικαίωμα επί τη βάση των κανόνων να απαντάτε μόνο σε μία από αυτές γιατί οι συνάδελφοι θα πρέπει να σεβαστούν τους κανόνες και δεν το κάνουν όλοι βέβαια. Οφείλουν να θέσουν μία ερώτηση στον χρόνο τον οποίο έχουν στη διάθεσή τους. Λίζιακ. Κυρία Άστον, η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπλέκεται σε πολλές διεθνείς σειράξεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Μία από τις προτεραιότητες της όμως θα πρέπει να είναι να προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αναφερθήκατε στα Βαλκάνια. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα τα οποία χαίνουν στη Γεωργία, της οποίας έχει παραβιαστεί η εδαφική ακαιρεότητα Υπάρχουν επίσης προβλήματα με τη Μολδαβία, ένα τμήμα της οποίας ε, ελέγχεται από αποσχιστικές ε, δυνάμεις στην υπερνηστερία κτλ. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ποια είναι η σχέση μας με τη Ρωσία γύρω από τα προβλήματα αυτά. Πώς μπορείτε να πείσετε τη Ρωσία να εγκαταλείψει αυτή την πολιτική διεύρυνση της ζώνης επιρροής της. Γκόμες ένα λεπτό. Πολλοί από εμά πιστεύουμε ότι αν δεν υπάρξει μια ουσιαστική αλλαγή από πλευράς του Ιράν, στη στάση των Ιρανών εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να φανούμε πάρα πολύ αυστηροί και να θέσουμε συγκεκριμένες κυρώσεις οι οποίες να είναι σωστά στοχευμένες και να θίξουν μόνο την κυβερνητική τάξη της χώρας αυτής. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει αυτούς οι οποίοι μάχονται για τη δημοκρατία και την ελευθερία στο Ιράν. για να σπάσει πια αυτό το σιδηρό παραπέτασμα το οποίο θέλει να επιβάλλει η θεοκρατική κυβέρνηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, δύο από τα σημαντικά νέα στοιχεία που έφερε η συνθήκη της Λισαβόνα στον τομέα της κοινή εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας είναι δύο ρήτρε. Να ξεκινήσετε από την αρχή παρακαλώ νέα στοιχεία που έφερε η συνθήκη της Λισαβόνας στον τομέα της κοινή εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας είναι δύο ρήτρε. Η ρήτρα αμοιβαία υποστήριξη, Mutual Assistance Clause, και η ρήτρα αλληλεγγύη, Solidarity Clause. Συγκεκριμένα η ρήτρα αμοιβαία υποστήριξη, το άρθρο 42.7 της συνθήκης, αναφέρει ότι αν ένα κράτος μέλος υποστεί στρατιωτική επίθεση στο έδαφο του, οι εταίροι του στην ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να του παράσχουν βοήθεια και υποστήριξη. Πώς αντιλαμβάνεστε την ουσία, το πνεύμα και την πρακτική αξία αυτού του άρθρου. Πιστεύετε ότι αυτή η ρήτρα αμοιβαία συνδρομής θα πρέπει και πώς να επηρεάζει τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών της και στην περίπτωση που μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ως επίσημη ξεκάθαρη και διακηρυγμένη πολιτική της την απειλή πολέμου κατά κράτους μέλους και δεν μιλάω θεωρητικά, η περίπτωση υπάρχει στα Νατιοανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. La replica alla signora vicepresidente per tre minuti. Την απάντηση θα δώσει η Αντιπρόεδρος μέσα σε τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ. Πρέπει να δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσονται τα θέματα αυτά στη Μολδαβία, στον Αγκόρνο Κάραμπαχ. Όπως είπα στην αρχή της ε, παρουσίασής μου, η πολιτική γειτονία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Καταρχάς στη Μολδαβία συνεργαστήκαμε, συνεργαζόμεθα μάλλον ε, σωστά, έχουμε Είμαστε η δεύτερη χώρα σε βοήθεια κατά κεφαλήν 60 ευρώ κατά πολίτη της χώρας προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον Αντμπόρνο Καραμπάχ γίνονται προσπάθειες και η Τουρκία στα πλαίσια της βελτίωσης των σχέσεων με την Αρμενία μπορεί να επηρεάσει και ε, φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις πραγματικότητες της περιοχής. Να δούμε λοιπόν ποια είναι τα θέματα αυτά, ποιες είναι οι σειράξεις και ποιες οι αιτίες. Η Ρωσία είναι θα έλεγα ένας κοινό παράγων ε, για πολλούς λόγους. Εμπλέκεται στην περιοχή αυτή, πολλές φορές εμπλέκεται θετικά στην περιοχή ε, και όταν πάω στην Μόσχα νομίζω θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μια θέση η οποία προληπτικά να αποβεί παραγωγική και χρήσιμη. Για την κυρία Γκόμες και σχετικά με το Ιράν και πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα είμαι σαφώς υπέρ ε, όλων των δράσεων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις σε αυτή τη φάση βέβαια για το που βρίσκεται τώρα πλέον το Ιράν. Οι κυρώσει φυσικά είναι μία οδός, θα δούμε το Συμβούλιο τι θα αποφασίσει, έχουν εκφράσει όμως την επιθυμία τους ότι θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος με βάση συγκεκριμένες αρχές όμως και να αναγνωρίσουμε ότι αν οι κανόνες δεν γίνονται σεβαστοί για ένα τέτοιο διάλογο θα πρέπει να αναλυφθεί δράσης. Σχετικά με την ρήτρα αλληλεγγύης. Έχω το 47-2 εδώ ανοιχτό μπροστά μου. είναι μια υποχρέωση και εφαρμόζεται έτσι και αλλιώς όπως ακριβώς και το 51 του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το εφαρμόσουμε αυτό. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει το Συμβούλιο, μια συζήτηση την οποία πρέπει να κάνει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, μιας και τώρα έχουμε τη συνθήκη στη διάθεσή μας, να δούμε ποιες είναι οι πρακτικές συνέπειες οι οποίες θα προέλθουν από το περιεχόμενο της συνθήκης. Η συνθήκη, αν θέλετε, προβλέπει μια γενική έκκληση, θα έλεγα, για υποστήριξη. Το θέμα είναι να δούμε και με ποιο τρόπο πιστεύει το Συμβούλιο θέλει να δώσει την ενέργεια την οποία έχει στη διάθεσή του προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα περνάμε στους προέδρους ή εκπροσώπους των προέδρων των συμμετεχουσών κοινοβουλευτικών επιτροπών. Κοινάδελφος Ζολή, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, Εξ ονόματος Επιτροπής Ανάπτυξης θα ήθελα να σας θέσω το ερώτημα για το ποιος επίτροπος θα είναι αρμόδιος για τον προγραμματισμό των δράσεων ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης και ποιος θα είναι ο ρόλος για τα θέματα ανάπτυξης της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων. Θα ήθελα επίσης να έχω παραδείγματα των συγκεκριμένων μέτρων που θα λάβετε για να εξασφαλίσετε το σεβασμό του άρθρου 208 της Συνθήκης Λισαβόνας που απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει υπόψη τους στόχους συνεργασίας και ανάπτυξης στην εφαρμογή πολιτικών που μπορεί δυνητικά να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες. Πώς θα εξασφαλίσετε λοιπόν την ενιαία δράση της εξωτερικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον σεβασμό αυτών των ρητρών. Επίσης, θα αντιταχθείτε στη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Κολομβία. Δύο λεπτά απάντησης από την κυρία Άστον. Για ένα ερώτημα βέβαια. Σας ευχαριστώ. Αλλάζουν οι κανόνες συνέχεια, βλέπω. Σε ό,τι αφορά τα θέματα ανάπτυξης. Θα ήθελα να σας πω ότι η ανάπτυξη βρίσκεται στην καρδιά του έργου το οποίο πρέπει να αναπτύξουμε στη σχέση μας με χώρες τρίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι συναρπαστικό το να βλέπουμε πως οι τρίτες χώρες χαίρονται ιδιαίτερα που εμείς προσπαθούμε να το πετύχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει πρέπει να αναγνωρίσουμε τη σημασία αυτής της πτυχής της πολιτικής. Και αυτό απαιτεί την προσοχή του Συμβουλίου αλλά και την Κομισιόν. Και ο κύριος Σπίμπαλξ που είναι υποψήφιος επίτροπος για τα θέματα αυτά έχει συνεργαστεί μαζί μου πάρα πολύ για το πώς μπορούμε να είμαστε αποτελεσματική. <clears throat> Ο στόχος μας είναι να υπάρχει και ένα γραφείο ανάπτυξης σε κάθε εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσικά για τα θέματα του ΕΤΑ είναι ο Επίτροπος Ανάπτυξης, ο οποίος παραμένει υπόλογο για τη διαχείρισή του, αλλά μέσα σε ένα στρατηγικό πλαίσιο προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε μια κοινή εξωτερική πολιτική. Είναι σημαντική λοιπόν η, η ανάπτυξη, παραμένει στα χέρια του Επιτρόπου Ανάπτυξης, αλλά θέλουμε να τη θέσουμε μέσα σε ένα συνεκτικό πλαίσιο. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι ένας πρακτικός τρόπος αντιμετώπισης που θα μας επιτρέψει να υλοποιήσουμε αυτό που έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο και χαίρομαι που ο Άντρες, Πίμπαλξ και εγώ θα συνεργαστούμε για το θέμα αυτό. Για τη Συμφωνία Ελευθέρων Εμπόριου με την Κολομβία. Πού βρισκόμαστε. Επειδή τώρα εγώ δεν είμαι πια επίτροπος εξωτερικού εμπορίου, από ό,τι γνωρίζω, φτάσαμε σε ένα σημείο των ε, διαπραγματεύσεων όπου αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να διακόψουμε αυτή τη διαδικασία διότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει την άποψή του βάσει τη συνθήκη τη Λισαβόνα για το θέμα αυτό και η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει υπόψη την άποψη του Κοινοβουλίου. Σε αυτή την ενδιάμεση λοιπόν φάση δεν έχει πολύ νόημα κατά την άποψή μα να προχωρήσουμε σε κάποια κατάληξη του διαλόγου. Δεν ξέρω αν συμφωνεί το Κοινοβούλιο. Κύριος Καζίνη Πρόεδρος της Συνταγματικής Επιτροπής για ένα λεπτό. Κύριε Άστον, μία απλή ερώτηση. Αν και βέβαια όταν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα η Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάσταση θα είναι πολύ περίπλοκη. Περιμένοντας το αίτημα του Συμβουλίου φυσικά. Στα πλαίσια των γραπτών απαντήσεών σας, ε, κύριε Αντιπρόεδρε, είπατε ότι η βασική σας προτεραιότητα είναι η δημιουργία της εξωτερικής υπηρεσίας, χρήσιμης, αποτελεσματικής, που θα το ζηλεύει ο κόσμος όλος. Πάρα πολύ ωραία. Σας ρωτάω λοιπόν. <clears throat> Μήπως θα πρέπει να δημιουργηθεί και μία ανωτάτη σχολή ευρωπαϊκής διπλωματίας, εκμεταλλευόμενη τις σχολές φυσικά που υπάρχουν στην Ευρώπη, έτσι ώστε να αποφυτούν νέοι από την σχολή αυτή, νέοι διπλωμάτες, οι οποίοι να γνωρίζουν πολύ καλά τη διπλωματική ιστορία της Ευρώπης και να είναι σωστά εκπαιδευμένοι στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων. Δύο λεπτά απάντηση η Αντιπρόεδρος Άστον. Τα πιο απλά ερωτήματα είναι και τα πιο ενδιαφέροντα πολλές φορές. Μπορεί να καταλήξουμε στο τέλος της θητείας μου σε μια φάση που θα έχουμε κάποιο σχήμα εκπαίδευσης για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Καταρχήν όμως θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτά που υπάρχουν ήδη παραδείγματος χάρη από την Κομισιόν η εκπαίδευση που δίνει στα άτομα τα οποία πηγαίνουν σε αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά τα οποία έχουμε από τα κράτη-μέλη για να διαμορφώσουμε ένα καθεστώς κατάρτισης που θα δώσει και στα άτομα που βρίσκονται τώρα στι αντιπροσωπείες κομισιών και στις υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν και για τους αντιπροσώπους των κρατών μελών τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να φέρουν σε πέρα στο έργο τους. Υπάρχει βέβαια μια σειρά επικρίσεων για το κατά πόσο είμαστε αποτελεσματικοί για την κατάρτιση. Το κολέγιο της Βρύγης είναι πολύ χρήσιμο για τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και τέτοια θέματα αλλά η εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας ιδιαίτερος φορέας. Θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη κατάρτιση των διπλωματών για να αναγνωρίσουν την ιδιοτυπία αυτού του νέου φορέα. Τώρα, πω, αν αυτό σημαίνει ενιαίο φορέα εκπαίδευση και κατάρτιση, αυτό δεν είμαι σίγουρη ακόμα ότι το έχουμε αποφασίσει. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών, κ. Στάσης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εδώ είμαι, εδώ είμαι κύριε Άστον. Οι συνάδελφοι Μπροκ και Νέτς έθεσαν ήδη σαφή ερωτήματα για αυτή την υπηρεσία εξωτερικής δράσης που θα είναι από τις μεγαλύτερες προτεραιότητές σας λοιπόν. Κατά την ακρόαση αυτή είπατε ήδη ότι Ποιος είναι ότι θα θέλατε να είστε υπόλογοι και να αναφέρετε τακτικά στο Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα της δράσης σας. Υπόσχεστε λοιπόν άρα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί να ασκήσει πλήρως τον ρόλο του δημοσιονομικού ελέγχου. Άρα η υπηρεσία αυτή εξωτερικής δράσης θα είναι μια χωριστή κατηγορία στον προϋπολογισμό και το Ελεκτικό συνέδριο θα μπορεί να την ελέγχει κανονικά η όλα θα μπορεί να παρέμβει, το κοινοβούλιο θα μπορεί να ελέγχει δημοσιονομικά τα πεπραγμένα της. Δύο λεπτά κυρία Άστον. Δύο λεπτά. Ελπίζω να μπορέσω να είμαι σύντομη γιατί νομίζω ότι είχα πει ήδη, είχα απαντήσει αυτό το ερώτημα προς τον κύριο Μπροκ. Υπάρχουν δύο τρόποι για να το δει κανεί. Μερικοί λένε ότι πρέπει να είναι τμήμα της Κομισιόν η υπηρεσία αυτή και άλλοι να είναι ξεχωριστή. Ό,τι και να γίνει, εγώ προτιμώ χωριστή, γιατί είναι σου generis υπηρεσία. Αλλά πάντως το Κοινοβούλιο θα μπορεί να παίξει τον ελεγκτικό του ρόλο, όποιος και να είναι τελικά, όποια να είναι τελικά η δομή της. Γιατί ο προϋπολογισμός της θα είναι τμήμα του γενικότερου προπολογισμού. Αυτό είναι φανερό. Και άρα θα είστε και εσείς συνυπεύθυνοι και για την απαλλαγή του. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν άρα είναι ποιο ρόλο θα παίζω εγώ στην απαλλαγή. Διότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι θα παίζουν το ρόλο που προβλέπουν οι συνθήκες και οι κανονισμοί, αλλά εγώ είμαι ανοιχτή για τις λεπτομέρειες. Πρέπει απλώς να δημιουργηθεί η δομή ώστε να υπάρξει και σωστή χρήση των κονδυλίων. Επίσης, ένα από τα σημαντικότερα θέματα είναι να υπάρχει αρκετή ευελιξία στον προϋπολογισμό της, όχι για να αποφευχθεί ο έλεγχος, αλλά για να αναγνωρίσουμε το γεγονός που διαπιστώσαμε πρόσφατα, δηλαδή ότι η κατάσταση αλλάζει πολύ γρηγορότερα από ό,τι προβλέπουμε. Δέστε τι έγινε με την Ιεμένη τις περασμένες εβδομάδες. Θα πάω και εγώ στη συνάντηση που θα συζητήσει το θέμα της Ιεμένης. Α, τέτοιου είδους θέματα δείχνουν ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα πολύ σύντομα και πρέπει να είναι ευέλικτος ο προϋπολογισμός. Αλλά το Κοινοβούλιο ούτως ή άλλως θα παίξει πλήρως το ελεγκτικό του ρόλο. Μορέιρα, πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αντικαθιστώ εδώ την κυρία Μουσκαρδίνη που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής μου και που είχε επιλεγεί για να την εκπροσωπήσει εδώ αλλά αναγκάζομαι να την αντικαταστήσω εγώ γιατί καθυστέρησε λόγω αεροπορικών συνθήκων. Κυρία Άστον μου, Γνωρίζετε ότι το εξωτερικό εμπόριο είναι σημαντικό τμήμα της πολιτικής της Ένωσης. Πώς προβλέπετε λοιπόν, πώς βλέπετε τον μελλοντικό σας ρόλο ως προς τον συντονισμό και τη συνεργασία με, τους καινούριους, με το καινούριο επίτροπο για το διεθνές εμπόριο. Δεύτερον, άλλο σημαντικό στοιχείο της νέα αυτής υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων είναι η μεταρρύθμιση των ε, ε, της εκπροσώπησης της Κομισιόν και της Ένωσης γενικότερα στο εξωτερικό οι οποίες μέχρι τώρα έχουν και ένα εμπορικό τμήμα εσείς πώς προβλέπετε την οργάνωση της εκπροσώπησης της Ένωσης της εμπορικής εκπροσώπησης της Ένωσης στα πλαίσια ή σε συνδυασμό με την εξωτερική αυτή υπηρεσία Είστε αποφασισμένοι να αποφύγετε διακυβερνητικές παρεμβάσεις στις εξωτερικές αυτές εκπροσωπήσεις. Α, με συγχωρείτε, αλλά θα σας διακόψω διότι πρέπει να σέβομαι τους χρόνους που έχουν προκαθοριστεί. Δύο λεπτά απάντηση από την κυρία Άστον. Εγώ προβλέπω να συνεργαστούμε σωστά και στενά. Είχαμε ήδη συζητήσεις για τον τρόπο της συνεργασίας. Το εμπόριο είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει να παραμείνει η κατάσταση αυτή ως έχει. Η σχέση φαίνεται ότι έχει εξελιχθεί καλά. Όταν εγώ επισκέφθηκα τις αντιπροσωπείες εκτός Ευρώπης σαν επίτροπος για το εξωτερικό εμπόριο, κατάλαβα ότι υπάρχει η δυνατότητα συλλογικής προσπάθειας και αποτελεσματικής προσπάθειας. Εγώ δεν θέλω να διαταράξω αυτή τη σχέση παρά μόνο εφόσον τη βελτιώσω. Δεν υποτιμώ βέβαια πόσο σημαντικό είναι το εμπόριο σχετικά με τα ευρύτερα στρατηγικά και οικονομικά μας συμφέροντα στον κόσμο. Το εμπόριο μπορεί να λειτουργήσει σαν κινητήρια δύναμη η οποία να δώσει την οικονομική στήριξη την οποία επιθυμούμε. Υπάρχουν χώρες με τις οποίες δεν έχουμε πολύ ισχυρέ ε, οικονομικές σχέσεις, εμπορικές σχέσεις, ε, όπως η Μολδαβία, αλλά προσπαθούμε να τις τονώσουμε μέσω της σύναψης συμφωνιών και με άλλες χώρες της περιοχής. Ε, νομίζω ότι πολλές χώρες θέλουν να ενισχύσουν τις εμπορικές τους σχέσεις μαζί μας και αυτά όλα θα καταστήσουν τις σχέσεις μας με τις χώρες αυτές στενότερες στο μέλλον. Νομίζω ότι θα συνεργαστώ σωστά με τον αρμόδιο επίτροπο για το εμπόριο, ο οποίος βέβαια θα παραμένει καθήλυν υπεύθυνο για τα θέματα αυτά. Επανερχόμεθα τώρα στις μεμονωμένες παρεμβάσεις βουλευτών ανά τρεις. Νόιζερ, ένα λεπτό παρακαλώ. <coughs> Κυρία Άστον, απαντώντας σε ένα ερώτημα για το Αφγανιστάν, είπατε ότι τα συγκεκριμένα αποτελέσματα θα πρέπει να ενισχύσουν την κατάσταση των ανθρώπων στο Αφγανιστάν. Εκεί έχετε την πλήρη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τουλάχιστον την ευρεία υποστήριξη. Η στοχοθεσία τώρα σε σχέση με την επικείμενη συνδιάσκεψη στο Λονδίνο για το Αφγανιστάν είναι σημαντική. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αποστολών και της εργασίας των ΜΚΟ στο Αφγανιστάν. Πώς θα συντονιστεί λοιπόν αυτή η προσπάθεια με το ΝΑΤΟ και το ΟΗΕ και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οι κοιό μπορούν να εργάζονται ανενόχλητοι και χωρίς την υποστήριξη των στρατιωτικών αρχών. Κύριο Σκέλαμ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Αστόν. Μετά από την ακρόασή σας το Δεκέμβριο, εγώ αποκόμισα την εντύπωση ότι οι κοινέ πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να βασιστούν σε υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες μεταξύ συμβαλωμένων μερών. Είσαστε σίγουροι ότι η εξωτερική μας πολιτική και η πολιτική ενέργεια μπορεί να βασιστεί σε συμφωνίες τύπου Πούτιν Σρέντερ, οι οποίες γίνονται και κλεισμένα των θυρών και πίσω από την πλάτη των κρατών μελών. Με ποιο τρόπο εσείς θα αποτρέψετε την επανάληψη τέτοιων διμερών συμφωνιών και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οι νέες συμφωνίες με τρίτες χώρες θα περιλαμβάνουν την ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προταθεί εδώ και πολύ καιρό από τον κύριο Σάρους Βόλς και εδώ και τρία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος Αλάκη για ένα λεπτό. εγώ θέλω να, να διαφωνήσω με τους ε, Βρετανούς συντηρητικούς συναδέλφους που σας κατηγορούν για τη θέση σας υπέρ της πυρηνικής, του πυρηνικού αφοπλισμού. Εγώ πάντα υποστήριζα ότι αυτό είναι το, καλύτερο κομμάτι του βιογραφικού σας <clears throat> και υποστηρίζω την στάση που είχε κρατήσει και ο κύριος Νταλέμα στο παρελθόν. Το ερώτημά μου είναι τώρα το εξή. Έχουμε τώρα μια ιστορική ευκαιρία. Σε λίγους μήνες θα γίνει η αναθεώρηση της συμφωνίας για τη διάδοση των πυρηνικών όπλων στα Ηνωμένα Έθνη. Μήπως θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ηγετικό ρόλο για τα πυρηνικά όπλα και την κατάργησή τους μετά από τις δηλώσεις του Πρόεδρου Ομπάμα. Κυρία Αντιπρόεδρε, έχετε τρία λεπτά να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Σχετικά για τη συνάντηση με το Αφγανιστάν και Νόιζα. 17 χώρες και οργανώσεις έχουν προσκληθεί να πάρουν μέρος στη συνάντηση αυτή και υπάρχουν και διαφορετικά θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Έχουν ήδη υπάρξει συναντήσεις με Αμερικανούς υπευθύνου. Ε, συναντήθηκα και με εκπροσώπους του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών και ένα από τα θέματα είναι να δούμε πώς θα συντονίσουμε καλύτερα τις παρεμβάσεις μας. Στόχος μας είναι να συντονιστούμε καλύτερα και να ενοποιήσουμε τις αντιπροσωπείες μας έτσι ώστε να μιλάμε με μία φωνή. Δεύτερον, να δούμε πόσο πιο αποτελεσματικοί μπορούμε να γίνουμε. Τι πρέπει να αλλάξουμε για να το πετύχουμε αυτό. Ας δούμε εκ νέου τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε. Ας εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις δυνατότητες συνεργασίας στο μέλλον. Για την ενεργειακή πολιτική. Όπως είπα προηγουμένως, απαιτείται να ακολουθηθεί μια ισχυρή πολιτική στον τομέα της διασφάλισης της προμήθειας ενέργειας. Αυτό σημαίνει πηγές ενέργειας, προέλευση ενέργειας, ήδη ενέργειας και αφορά επίσης και το τι θα κάνουμε με την ενέργεια την οποία εισάγει γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις, πάρα πολλοί αγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου που προτείνονται και που βρίσκονται σε στάδιο εγκατάστασης ή προγραμματισμού τώρα. Απαιτείται λοιπόν να υπάρξει μια συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας και θα συνεργαστώ με τον αρμόδιο επίτροπο για την ενέργεια για να το πετύχουμε σχετικά με τη, με τη συνθήκη διάδοσης. Ε, ξέρετε ότι σχετικά με, την με τον μονομερή αφοπλισμό το θέμα είναι το εξής. Θα πρέπει να προσπαθούμε να δούμε με διαφορετικό τρόπο τα πυρηνικά όπλα σήμερα. Να δούμε αυτά τα οποία έχει πει ο πρόεδρος Ομπάμα που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ξεκάθαρες απόψεις και θα πρέπει να τις συνδυάσουμε. Όπως και όλοι που βρίσκονται εδώ σήμερα, πιστεύω και εγώ ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά, τα οποία παρουσιάζουν τεράστιους κινδύνους για το μέλλον. Ιδιαίτερα όταν βλέπουμε το τι συμβαίνει ε, σε κάποιες ε, χώρες όπως το Ιράν και όπως ε, η έλλειψη ασφάλειας γύρω από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και τα προβλήματα τα οποία στοιχειοθετεί η τρομοκρατική απειλή. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε λοιπόν. Με ενδιαφέρουν τα θέματα αυτά και θα προσπαθήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τα προωθήσω σε συνεργασία φυσικά στενή με εσάς. φέρε ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, έχετε τονίσει από τότε που έχετε αναλάβει τα καθήκοντά σας τη σημασία του διατλαντικού διαλόγου. Εντάξει, αλλά Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα σχέδια, υπάρχουν προτεραιότητες, υπάρχουν θεσμικά εργαλεία σε αυτό το διατλαντικό διάλογο. Σε μια μελέτη ενός αμερικανικού think tank αναφέρεται ότι χάνεται ο κόσμος ο οποίος οδήγησε στη διατλαντική ε, συνεργασία. Η Αμερική και η Ευρώπη θα πρέπει να αναμορφώσουν με πιο αποτελεσματικό και στρατηγικό τρόπο τη σχέση τους και να την κάνουν μια εταιρική σχέση. Τώρα, τη στιγμή που έχουμε διαφορές με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραγωγικά το ρόλο των ανθρωπινών δικαιωμάτων για την παγκόσμια διακυβέρνηση ή τα θέματα τροφοδοσίας ενέργειας ή κλιματικής αλλαγής. Ποια είναι τα σχέδια προτεραιότητας και οι στρατηγικοί στόχοι που εσείς θα επιλέγατε για την αναμόρφωση των διατλαντικών σχέσεων. Ζημάνσκι για ένα λεπτό. Κύριε Αντιπρόεδρε, εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Αναφέρατε το ζωτικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ένωση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεθνώ. Και ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα τα οποία παραβιάζεται όλο και συχνότερα είναι η θρησκευτική ελευθερία. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια συμβάντα. Συνήθως αιματηρά στην Αίγυπτο και στο Βιετνάμ και στο Πακιστάν όπου ε, γίνονται επιθέσεις κατά χριστιανών ακόμη και στη Δημοκρατική Ινδία. Και υπάρχουν περιορισμοί των δυτικών χριστιανικών δογμάτων που εφαρμόζονται στην Κίνα και στην Ρωσία. Τι θα κάνετε λοιπόν για να αλλάξει η κατάσταση αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τελείως. Δεν λέει απολύτως τίποτα για την, τους διωγμούς των χριστιανών διεθνώς. Κόβατσεφ για ένα ολόκληρο λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Άστον. Εδώ, εδώ. Μας απογοητεύσατε όταν είπατε ότι δεν είστε πεπισμένοι για την ανάγκη ακροάσεων για τις υψηλές διπλωματικές θέσεις διότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα και μακρόσυρτη. Για να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και να είναι όλοι υπόλογοι ως, και ιδίω αυτοί οι εκπρόσωποι στις εξωτερικές υπηρεσίες τουλάχιστον στις αρμόδιες επιτροπές θα μπορούσατε να οργανώσετε οργανώσει ιδίω για σημαντικές ε, εκπροσωπήσεις όπως τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα κτλ. Ελπίζω να υποβάλλετε τη σχετική πρόταση αργότερα μέσα στο χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αντιπρόεδρε για τρία λεπτά. και πάλι ευχαριστώ για τις ερωτήσεις για την πολιτική μας έναντι τον ΗΠΑ έχετε δίκιο ότι πρέπει να πούμε ότι υπάρχει δυνατότητα να εξετάσουμε πόσο αποτελεσματικές είναι οι στρατηγικές μας σχέσεις με τα ΗΠΑ. Έχουμε εργαλεία και οργανωμένους διαλόγους στο Συμβούλιο Ενεργείας και άλλα. Και ιδίως από την πλευρά της Κομισιόν γίνονται τακτικές συναντήσεις με υπάτους εκπροσώπους τον ΙΠΑ. Νομίζω όμως ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα και δεν ξέρουμε ακόμη ποια ακριβώς εργαλεία διαθέτω. Είναι σαφές όμως ότι πρέπει να ενδυναμωθεί η σχέση που έχουμε στο δικό μου τουλάχιστον επίπεδο έτσι ώστε η Προεδρία του Συμβουλίου και της Κομισιόν να μπορεί να είναι πιο συντονισμένη. Ένα παράδειγμα από την εμπορική μου ζωή είναι οι συνεννοήσεις για τις εμπορικές διευκολύνσεις με αφρικανικές χώρες, όπου κοινό ήταν ο στόχος μας με τα ΣΥΠΑ. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν λοιπόν και έχετε δίκιο που το τονίζετε. Για τη θρησκευτική ελευθερία, η Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη χώρα που γνωρίζω, τη δική μου δηλαδή, σημαίνει σαφώς και θρησκευτικές ελευθερίες και για μένα είναι απολύτως τμήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λυπούμε που θεωρείτε ότι η Ένωση σιώπησε λέτε από αυτού, αλλά είναι προφανές ότι πρέπει, δεν πρέπει να το χωρίσουμε από άλλα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, για τους εκπροσώπους, εξωτερικούς εκπροσώπους. Και πάλι λυπούμε που σας απογοήτευσα, αλλά πρέπει να μπορώ να αποδείξω ότι έχω ορίσει τους καταλληλότερους. Δεν είμαι κατά των ακροάσεων στο Κοινοβούλιο, απλώς δεν είμαι πεπισμένη ότι το να καλούνται εδώ και να ακολουθείτε αυτή η μακρόσυρτη διαδικασία είναι το καλύτερο, διότι πρέπει να βρούμε κάποια άλλη μέθοδο όπου να σας ικανοποιεί και εσάς ότι είναι κατάλληλος ο διοριζόμενος. Θα το σκεφτώ, θα το σκεφτώ. Ο κύριος Σίγουιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ίσως ζητάμε πολλά, αλλά και εσείς απαντάτε πολύ γενικόλογα πρέπει να σας πω. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αμφότερη μία από πιο αληθινή γλώσσα. Την επομένη των εκλογών στην Ουκρανία υπάρχει καμία πρόθεση της Ένωσης για κάποια αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας αυτής. Γιατί στο Ουκρανία αντιμετωπίζουμε πολιτικό χάος. Και αυτό βολεύει πολλούς Ευρωπαίους. Να μην κάνουν τίποτε για την Ουκρανία δηλαδή. Υπάρχει μήπως καμία πρόθεση να σταματήσουν οι διαδικασίες σύνδεσης, να σταματήσουν οι συνεννοήσεις για τη διευκολύνση των θεωρήσεων. Σε ένα ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφρασε την άποψή του για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες λέγοντας ότι ήταν η πιο σημαντική στρατηγική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ψήφισμα αυτό είχε συγκεκριμένες προτάσεις για μηχανισμούς και εργαλεία βελτιωμένα για να ενισχυθεί αυτή η σχέση. Παραδείγματος χάρη δύο σύνοδοι κορυφή το χρόνο και όχι μία μονάχα και δημιουργία ενός διατλαντικού συμβουλίου όπου θα μπορείτε και εσείς να λαμβάνετε ε, μέρος μαζί με την κυρία Κλίντον. Επομένως, συμπλήρωση των εργαλείων που υπάρχουν ήδη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να προωθήσουμε την διατλαντική αγορά που αναφέραμε προηγουμένως και επίσης ένα ενεργειακό συμβούλιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι πιστεύετε όμως για αυτές τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δύο ε, συνοδικορφή του χρόνου και ένα συμβούλιο. Η κυρία Πακ. Εξ ονόματος του κυρίου Πόσελ θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Με ικανοποίησε η απάντησή σας ότι θέλουμε να έχουμε μια Ευρώπη που μιλάει με μια φωνή και που έχει συνεκτικότητα. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει στο παρελθόν. Το παράδειγμα του Κωσφοπεδίου δείχνει την κακοφωνία μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μας δείξετε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε μία ενιαία κατεύθυνση και σε μία μοναδική φωνή. Έχετε το λόγο κυρία ε, Πίτροπε, για, ένα, για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Σίβιατς. Δεν προσπάθησα να φανώ υπερβολικά πολιτικά ορθή ούτε γενικόλογη. Παρ' όλα αυτά κατανοείτε ότι καθώς αναπτύσσω τη στρατηγική μου και τα προγράμματα που έχω στην αυτή τη στιγμή έχω ξεκινήσει, πρέπει να μιλώ προσεκτικά για τα θέματα αυτά. Για την Ουκρανία σαν παράδειγμα. 17 Ιανουαρίου έχουν εκλογές τον πρώτο γύρο και τον Φεβρουάριο θα ακολουθήσει ο δεύτερος γύρος. Κανένας δεν γνωρίζει ποιος θα είναι ο νικητής της εκλογικής διαδικασίας και αυτό ίσως να αποδεικνύει το ότι λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα αυτή. Μετά τις εκλογές δύο στόχους πρέπει να έχουμε. Πρώτον, ποια θα είναι η σχέση με τη Ρωσία, ανάλογα με το ποιος θα νικήσει στις εκλογές. Πώς θα υποστηρίξουμε εμείς την Ουκρανία σε τομείς με τους οποίους έχουμε ήδη συνεργαστεί μέχρι τώρα. Σαν παράδειγμα η αποκατάσταση του δικαστικού συστήματος της χώρας. Έχουμε πάρα πολλή δουλειά επίσης στον τομέα του εμπορίου. Έχουμε ξεκινήσει τη δουλειά αυτή, αλλά υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος. Συνεπώς δεν είναι ότι εγώ δεν έχω ξεκάθαρες εικόνες για τους τομείς τους οποίους συζητάμε τώρα. Θα πρέπει να είμαστε όμως υπομονητικοί μέχρι την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και να μην προκαταλάβουμε τις συζητήσεις που θα έχουμε με τους Ικρανούς μετά. Σχετικά με τις ΗΠΑ Πολιτείες είπαμε ήδη πολλά. Είχα ήδη μια επαφή με την Υπουργό Εξωτερικών, την Χίλαρη Κλίντον, συναντηθήκαμε, Έχουμε προβλέψει επίσης και μία συνάντηση σύντομα στη Washington. Ήδη μίλησα μαζί της τηλεφωνικά και θα συναντηθούμε εκ νέου όταν ε, έχουμε αυτή τη δυνατότητα σύντομα. Πρέπει να ενισχύσουμε τον πολιτικό διάλογο και ένα από τα θέματα στα πλαίσια του οικονομικού και πολιτικού διαλόγου είναι να προωθήσουμε και την διακοινοβουλευτική συνεργασία με τη ΣΥΠΑ. Εγώ σαν επίτροπος εμπορίου, υπεύθυνη για το εμπόριο, συναντήθηκα με πάρα πολλά μέλη ε, του Κογκρέσου των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί γνωρίζουμε το ρόλο που παίζει στο Αμερικανικό σύστημα διακυβέρνησης. Ελπίζω και οι να αναγνωρίσουν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να υπάρξει ένας ισχυρότερος διάλογος στο μέλλον ανάμεσα στα νομοθετικά σχέλη ε, των εξουσιών της κάθε χώρας. Σε ευχαριστώ για τις ευχές της κυρίας ΠΑΚ. Ξέρετε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για τις χώρες που δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία του κοσφοπεδίου. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ο τομέας Γιούλεξ, ο οποίος λειτουργεί σωστά, αρκετά σωστά. Συνεπώς, είμαι πραγματίστρια σε σχέση με τι μπορώ να πετύχω, τουλάχιστον βραχοπρόθεσμα. Αλλά πάντως το θέμα είναι ότι το Γιούλεξ μπορεί να βοηθήσει σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη ή Μούνιτς. Κυρία, ευχαριστώ. Αναφερθήκατε στην Κούβα κυρία Άστον και στην Κολομβία. Η στρατηγική σχέση μεταξύ Ένωσης και Λατινικής Αμερικής ξεπερνάει βέβαια τις δύο αυτές χώρες και προβλέπονται πολλές διασκέψεις κορυφής για τη Χιλή, την Αργεντινή, ένα σχέδιο δράσης που να καθορίζει τους τρόπους εφαρμογής του διαλόγου με την Ήπειρο αυτή. Σύμφωνα με την εντολή σας λοιπόν, τι αξία δίνεται στη συνεργασία με τη Λατινική Αμερική πέρα από τις μεμονωμένες περιπτώσεις των δύο αυτών χωρών και τις εμπορικές σχέσεις. Επόμενο ευχαριστώ. Πριν από καμιά ώρα, κυρία Άστον, είχατε πει απαντώντας στην κυρία Χάουταλα Εμένα με ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα, τα απτά αποτελέσματα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αλλά η εξωτερική πολιτική αντιμετωπίζει συνεχώς διλήμματα. Είναι φυσικό, παραδείγματος χάρη. Ένας από τους στρατηγικούς εταίρους της Ένωσης ξέρουμε ότι εκτελεί συνεχώς ανθρώπους ή δολοφονεί δημοσιογράφους. Ποια λοιπόν θα είναι η προτεραιότητά σας, τα εμπορικά ή τα ανθρώπινα δικαιώματα. κύριος Γιάτεν Μάκιν Κυρία Μάκη. Κυρία Επίτροπε, η Λισαβόνα, η συνθήκη της Λισαβόνας έχει σαν στόχο να προωθήσει την ειρήνη στον περίγυρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευμάρεια για όλους. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πράγματι εξασφαλίσει αυτά τα πράγματα για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αλλά δυστυχώς η πρόληψη της βίας και των συγκρούσεων δεν βρίσκονται ακόμα στην καρδιά της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιζητήσει ένα νέο ρόλο ως ως ε, συμφιλιωτής και ως προαγωγός της ε, ειρήνης στον κόσμο. Τρία λεπτά για την κυρία Άστον. Ευχαριστώ για τη Λατινική Αμερική. Ναι, σύμφωνο είναι πολλά τα οποία μπορούν να γίνουν. Ε. Θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα για τη σχέση μας με την Λατινική Αμερική και υπάρχει ήδη πολύ ενδιαφέρον από την πλευρά της Ισπανικής Προεδρίας για την Λατινική Αμερική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τους επιτρόπους οι οποίοι ασχολούνται με περιφερειακές πτυχές. Ο στόχος του να έχουμε μια τέτοια κατανομή καθηκόντων δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε για μεμονωμένες χώρες. Πολλές φορές όμως οι χώρες λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο σαν ενότητες. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μια περιφερειακή στρατηγική και αυτό προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε και βασιζόμαστε και στις προτάσεις των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά τα οικονομικά δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση. Είναι θεμελιώδη τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι η θεμέλη λύθη της πολιτικής μας, αλλά και οι οικονομικές σχέσεις είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των σχέσεων με όλες τις χώρες του κόσμου. Έχουμε τις αξίες μας, τις θέσεις μας, θέλουμε να είναι σαφείς και ορατές οι αξίες μας. Αλλά θέλουμε να υπάρξει και ανάπτυξη και σε άλλες χώρες για να μπορέσουν να συνεργαστούν μαζί μας σε θέματα που μας ενδιαφέρουν. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, πρέπει να καλύψουμε και τις δύο πτυχές. Σε σχέση με αυτά που η κυρία Γιάχτεμακή. Θα σας πω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε όχι μόνο τη διατήρηση της ειρήνης, αλλά την επίτευξη και τη δημιουργία της ειρήνης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα Ηνωμένα Έθνη. Να εστιάσουμε την προσοχή μας στο πώς θα μπορέσουμε να προαγάγουμε την επίτευξη της ειρήνης και την αποφυγή των συγκρούσεων. Ένα θέμα το οποίο εμένα με οδήγησε σε μεγάλη συνειδητοποίηση μετά από την συνδιάσκεψη Κοπενχάγης. Βλέποντας πολλές από τις εκθέσεις για τη σταθερότητα σε όλο τον κόσμο, είναι φανερό ότι υπάρχουν πολλά κράτη τα οποία αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα λόγω της κλιματικής αλλαγής και θα αντιμετωπίσουν και στο μέλλον, γιατί άμεσα ή έμεσα θα δημιουργήσει προβλήματα ακόμα και χάος στις χώρες αυτές η κλιματική αλλαγή και θα οδηγήσει σε δυνητικές συγκρούσεις. Κάτι λοιπόν το οποίο πρέπει να δούμε για το ρόλο μας στον κόσμο είναι πώς θα εξασφαλίσουμε την απαραίτητη σταθερότητα για να αντιμετωπίσουμε θέματα τέτοιου πλανητικού χαρακτήρα. Ένα παράδειγμα λοιπόν μονάχα σας δίνω όπου η οικοδόμηση της ειρήνης η δυνατότητα να έχουν οι χώρες αυτές την υποστήριξη που θέλουμε που βασίζεται σε απόψεις μας και τις αξίες μας να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά για να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές οικονομικά, πολιτικά, ακόμα και στρατιωτικά είναι δυνατό, αλλά για να επιληθούν τα προβλήματά τους. Αν το κάνουμε αυτό θα έχουμε πράγματι επιτύχει τους στόχους μας. Ζάλα, ένα λεπτό πρέπει να μην ξεχνάμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξέρετε ότι έδωσε το βραβείο Σαχάροφ στην ρωσική οργάνωση, στη ρωσική ΜΚΟ Memorial. Για μια ακόμη φορά έχουν παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ρώσων πολιτών. Και ένας από τους εκπροσώπους της οργάνωσης Memorial έχει πλέον είναι στη φυλακή μάλλον. Λοιπόν, πώς ακριβώς εσείς θα αντιμετωπίσετε την υποβόσκουσα αντίφαση ανάμεσα στις αξίες από τη μία στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς όπως ε, η ενέργεια, η ασφάλεια, το Ιράν κτλ. Πώς θα διαχειριστείτε τις αντιφάσεις αυτές. Εμείς δεν θέλουμε να διώξουμε τη Ρωσία από τις ευρωπαϊκές αξίες, θέλουμε να τη φέρουμε πιο κοντά μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρομαι στους εταίρους μας προς Ανατολάς, ιδιαίτερα τη Λευκορωσία και τη Ρωσία. Pytanie, jaka polityka wobec Białorusi, w której ciągle mamy do czynienia z więźniami. Όταν είχα θέσει ένα ερώτημα παλαιότερα μου είχατε πει ότι θα μου απαντήσετε σε υστερότερη φάση. Ιδιαίτερα στη Λευκορωσία τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται σε καμία περίπτωση σεβαστά. Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι ώστε να υπάρξουν αλλαγές στη Λευκορωσία. Μπορούμε να πιέσουμε μέσω των οικονομικών σχέσεων ή τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν αντιμετωπίζονται με τον πιο σοβαρό τρόπο. Το ίδιο ισχύει και με την Κούβα. Θέλετε εσείς να ακολουθήσουμε την άποψη της Ισπανικής Προεδρίας ή πιστεύετε ότι υπάρχει διαφορετικός τρόπος για την αντιμετώπιση των σχέσεων με την Κούβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε έχουμε το θέμα της Ερυθρέας, η οποία έχει προβλήματα με την ε, λειτουργία των αστυνομικών της δυνάμεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προσπαθήσει στο παρελθόν να βοηθήσει στην ανάπτυξη καροτήτων την ε, Ερυθρέα και έχουν δοθεί σημαντικά κονδύλια προς την κατεύθυνση αυτή. Αναρωτιέμαι κυρία Άστον αν θα χρησιμοποιήσετε αυτό το διάβλο επιρροής προς την Ερυθρέα για να τους ζητήσετε να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί υπάρχουν πολλοί δημοσιογράφοι οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή στην Ερυθρέα και είναι άγνωστοι η τύχη τους πολλές φορές. Μπορεί να είναι μικρή αυτή η χώρα, αλλά είναι σημαντικό και σε αυτή την συγκεκριμένη περίπτωση να ξέρουμε πώς θα προσπαθήσετε εσείς να ασκήσετε πίεση και να χρησιμοποιήσετε το μοχλό της ε, βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βελτιώσετε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για να μπορέσει η Ερυθρέα να εγκαταλείψει αυτές τις αποτρόπες μεθόδους που χρησιμοποιεί η κυρία ε, Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για τρία λεπτά για να απαντήσει. Κυρία Τζάλα, δεν ήξερα για τη σύλληψη αυτή που αναφέρατε. Νομίζω ότι το ερώτημα δεν είναι τι θα κάνω εγώ, αλλά τι θα κάνουμε εμείς. Γιατί ξέρω ότι όταν προσπαθούμε να υποστηρίξουμε φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει να διαδραματίσει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, προφανώ. Αλλά όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να αναπτύξουμε από κοινού. Το ερώτημα είναι τι στρατηγική να αναπτύξουμε για το μέλλον. Να βασιστούμε σε αυτά που ήταν επιτυχή στο παρελθόν, αλλά και να ανασκευάσουμε αυτά τα οποία δεν λειτουργήσαν. Εγώ δεν έχω λοιπόν συγκεκριμένη λύση προς το παρόν. Αυτό το οποίο έχω να υπάρχει, την, ε, έχω την συνειδητοποίηση ότι χρειάζεται μια α, σαφήνεια για τα θέματα αυτά. Για τη Λευκορωσία ίσως δεν έχω απαντήσει πλήρως, αλλά εν ώψη των εκλογών του 2010 και του 2011 είναι μια πολύ σημαντική χώρα η Μπελαρούς. έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την ε, Τελωνιακή Ένωση που θέλει να οικοδομήσει η Ρωσία με την Πελαρούς, τη στρατηγική αυτή σχέση και τις συνέπειες οι οποίες θα προκύψουν. Ξεκινήσαμε τον Ιούνιο στην Πράγα τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Λευκορωσία. Ήταν ενδιαφέρον αυτό, αλλά δεν έχω ακόμα κάποια στοιχεία ανάδρασης για να ξέρω προς τα που θα κινηθούμε. Είναι πολύ θετικό ότι ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση με την Πελαρούς. Χρειαζόμαστε όμως να εξασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η απαγόρευση χορήγησης προξενικών θεωρήσεων και να υπάρξει πραγματικά πίεση για φιλελευθεροποίηση μέσω αυτού του εργαλείου στην Μπελαρούς. Και φυσικά πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει με τη στάση της Ρωσίας για την Τελωνιακή Ένωση με την Μπελαρούς, τη Λευκορωσία. Όλα αυτά σιγά σιγά είναι ψηφίδες του παζλ το οποίο αρχίζει πια να συγκροτείται. Με ρωτήσατε και για την Κούβα. <clears throat> Εκεί έχουμε μια πάρα πολύ σαφή πολιτική και μονάχα με ομοφωνία μπορεί να αλλάξει το Συμβούλιο τη θέση του. Αυτή είναι η πολιτική που ακολουθήθηκε εδώ και 13, κράτη, 13 χρόνια. Πολλά κράτη-μέλη έχουν ανησυχήσει και πάλι για τα ζητήματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το μόνο θέμα το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι το να δούμε αν υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε οι αλλαγέ που μπορούμε να επιφέρουμε στις πολιτικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είμαστε το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί. Και γι' αυτό το ερώτημα είναι αν ήταν αποτελεσματική αυτή η πολιτική μας για τα τελευταία 13 χρόνια και αν το Συμβούλιο θέλει να αλλάξει. Μέχρι τότε η πολιτική μας παραμένει. Ξέχασα, ξέχασα, ξέχασα για την κυρία Σβένσον και την Ερυθρέα. Το θέμα της αστυνομικών δυνάμεων. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, αλλά η αρχή αυτή που αναφέρατε σε σχέση με την χρήση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πίεση που θα πρέπει να ε, εφαρμοστεί για την ελευθερία του τύπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό τονίζω ότι έχουμε μια σημαντική πολιτική άποψη για τα θέματα αυτά Μπορούμε να παίξουμε και ρόλο σε οικονομικό ακόμα και σε στρατιωτικό επίπεδο και για όλα αυτά είναι σημαντική ερυθρέα. Κούκαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας Λέβη Άστον. Το ερώτημά μου αφορά την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων που είναι πολύ σημαντική για τη μελλοντική διεύρυνση της Ένωσης. Αναφέρατε σύντομα στην αρχική σας εισήγηση και απαντώντας στον κύριο Γιώκο Κάτσεν ορισμένα πράγματα, αλλά θα ήθελα να μας πείτε ποιος θα ήταν, ποια θα ήταν τα αποτελεσματικότερα μέτρα της Ένωσης για να ενταχθούν οι χώρες αυτές στην Ένωση έτσι ώστε να ενδυναμώσει την Ευρώπη η ένταξη αυτή. Και ποιο ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα προβλέπετε για την λήξη των ενταξιακών διαδικασιών και τι και αν προβλέπετε να κάνετε στα πλαίσια της εξωτερικής υπηρεσίας. Γκουαλτιέρη. Ανάμεσα στις προτεραιότητες δεν άκουσα τη Σομαλία, ένα δραματικό θέατρο κρίσης, μια σύραξη πάρα πολύ σοβαρή. Έχουν ξεκινήσει επίσης και μάχες με την Αιθιοπία στη Μεθόριο και έχουμε μια θα έλεγα σημαντική στρατιωτική ε, παρουσία εκεί. Ε, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε ε, την στρατιωτικές δυνάμεις της Σομαλίας ή θα θέλαμε τουλάχιστον όπως επίσης και την ακτοφυλακή της χώρας αυτής. Τι προοπτικές έχουμε. Η τελευταία τροπολογία στην οποία κατέληξε ε, το Συμβούλιο για την Αποστολή Αταλάντα σχετικά με την παρακολούθηση των αλλιευτικών δραστηριοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι θα προστατευθούν και τα ευρωπαϊκά αλλιευτικά σκάφη ή απλά θα ελεγχθεί η παράνομη αλλιευτική δραστηριότητα. Απάντηση της κυρίας Άστον τρία λεπτά. Um, uh, Δύο ερωτήματα, έτσι δεν είναι. Για να μην κάνω λάθος. Για τα Δυτικά Βαλκάνια. Νομίζω ότι η αποτίμηση της, στην οποία έχουμε προβεί μας λέει ότι το μέλλον τους βρίσκεται στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευκαιρία να γίνουν τμήμα του μέλλοντος της Ευρώπης. Για κάποιες χώρες στην περιοχή αυτή ήδη είναι εν εξελίξει αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν χώρε με τι οποίε είμαστε, οι οποίες είναι έτοιμε να ξεκινήσουν διάλογο και για τι οποίε έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα προχωρήσουμε. Εστίασα προηγουμένως στη Βοσνία γιατί ανησυχώ ιδιαίτερα για το πρόβλημα αυτό και το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που λαμβάνουν χώρα εκεί. Εκεί χρειάζεται ευρύτερο διάλογο για να πετύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Γιατί έχουν περάσει 13 χρόνια από τη Συμφωνία Dayton και οι κύριοι εμπλεκόμενοι δύο συνομένες Πολιτείες ξέρετε ότι εξακολουθούν να έχουν το κλειδί. Ο Καρλ κατά την Σουηδική Προεδρία είχε πολλές επαφές με τους Αμερικανούς. Μπορώ να σας απαντήσω μονάχα γενικά, γιατί βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου θα πρέπει να δούμε αν αυτή η διαδικασία το λεγόμενη των 5 συν 2 είναι αποτελεσματική, αν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα. Σίγουρα όμως το, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι μια χώρα όπου απολαμβάνουν σεβασμού όλες οι εθνοτικές ομάδες και η οποία μπορεί να προχωρήσει σε οικονομική ανάπτυξη και το χρονικό πλαίσιο του, της επίτευξης αυτού του στόχου πρέπει να είναι ορατό. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε στο επίπεδο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μόναχα. Τώρα πώς ακριβώς θα γίνει αυτό. Δεν γνωρίζουμε μέχρι να ακούσουμε την απόψη των εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων. Και εδώ φυσικά θα παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αναπτύξει αυτή τη δυναμική με μια ενιαία φωνή στην περιοχή, ιδίω στη Βοσνία όπου εμπλέκονται χώρες όπω η Ρωσία, η Τουρκία, οι Ηνωμένες Για τη Σομαλία <clears throat> θα πρέπει να ενισχύσουμε την Αταλάντα. Λαμβάνω υπόψη αυτό το οποίο λέτε για την παράνομη αλία. Δεν γνωρίζω τα θέματα αυτά. Το ερώτημα του μέχρι ποιου σημείου μπορούν να διακριβώσουν τι ακριβώς κάνει ο καθένας η Αταλάντα δεν το ξέρω, αλλά είναι μια πολύ αποτελεσματική και σημαντική ε, αποστολή και είναι σημαντικό να μπορούμε να συλλαμβάνουμε τους πειρατές και να τους διώκουμε και κάνουμε προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. Πρέπει να σκεφτούμε όμως τι θα κάνουμε και στο έδαφος της Σομαλίας, γιατί δεν αρκεί η αστυνόμευση των θαλασσών, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε προγράμματα εκπαίδευσης που συζητούνται από την Επιτροπή Ντάρτμουτ για ένα λεπτό. Ήσασταν μία από τους τέσσερις υπαλλήλους του CND της ε, οργάνωσης ε, κατά, της, κατά των πυρηνικών όπλων. Ήσασταν ε, μία από τους τέσσερις που παίρνατε μισθό θα έλεγα. Αν οι απόψεις σας και οι φίλοι σας του CND είχαν επικρατήσει, η Ανατολική Ευρώπη δεν θα ήταν ελεύθερη πλέον. Στην πιο σημαντική και στο πιο σημαντικό πρόβλημα στις εξωτερικές μας υποθέσεις η άποψή σας ήταν δυστυχώς λανθασμένη. Είστε η Εντίθ Πιάφ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πείτε κι εσείς το «Rien de rien, je ne regrette rien». Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσετε συγνώμη από όλους αυτούς τους οποίους στο παρελθόν παραπλανήσατε. Δύο λεπτά η υποψηφία. Όχι, όχι, δεν φοβάμαι καθόλου να απαντήσω. Απλά περίμενα ερωτήσεις σχετικές με τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. μπορείτε τα θέματα αυτά να τα συζητήσετε όπως θέλετε στα πλαίσια της γενοβουλευτικής δημοκρατίας. Έχουμε 27 χώρες οι οποίες είναι παρούσες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακριβώς στα πλαίσια της δημοκρατίας και της χαράς που νιώθω που συμμετέχω στις δημοκρατικές διαδικασίες. Όλα αυτά είναι γνωστά αυτά που είπατε, είναι γνωστά ανέκαθεν. Ναι, Προφανώς οι απόψεις αλλάζουν με τα χρόνια, βλέπετε ακριβώς ε, ε, το ότι δεν έχω κρύψει ποτέ την, ε, τις δουλειές, τις θέσεις εργασίας τις οποίες είχα μέχρι τώρα. Εγώ διαδήλωνα γιατί πίστευα ε, για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Μπορείτε να λέτε ότι δεν το επεδίωκα με τον σωστό τρόπο ίσως, αλλά παρόλα αυτά Είχαμε σχέσεις και με, τα, με τις ομάδες ε, οι οποίες έκαναν αντίσταση στην Ανατολική Ευρώπη τότε. Ε, δεν φοβόμασταν την Ευρώπη εμείς τότε, θέλαμε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα και οι αξίες τις οποίες πάντα υποστήριξα είναι αξίες ε, τις οποίες, στις οποίες βασίζεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα λεπτό Σόλτς. Κυρία Υποψήφια, κύριε Πρόεδρε, αντίθετα από τον κύριο Τάνοκ, μπορώ να σας πω ότι χαίρομαι πραγματικά που είχατε αυτή την νεανική όρμη στα νιάτα σας για, την, ε, για τον μονομερή αφοπλισμό. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα θέματα αυτά των πυρηνικών όπλων είναι ένα από τα συγκεκριμένα ζητήματα που σας ενδιαφέρει και εδώ θα ήθελα να σας θέσω το ερώτημα με ποιο τρόπο μπορεί να προχωρήσει η διάσκεψη για την επαλήθευση και την ε, μη περαιτέρω διασπορά των πυρηνικών όπλων και να μην έχει τα ίδια αποτελέσματα με την διάσκεψη της Κοπενχάγης. Γιατί όλα αυτά, όλες αυτές οι αποτυχίες είναι αποτυχίες για την πολιτική και τελικά αποτρέπουν τα άτομα από το να λαμβάνουν μέρος στην πολιτική. Λοιπόν, η διάσκεψη αυτή για την επαλήθευση θα πρέπει να έχει αποτελέσματα και ποια είναι τα συγκεκριμένα σχέδια τα οποία μπορείτε εσείς να κατανομάσετε τα οποία μπορούν να επιτύχουν μέσα σε αυτήν την διάσκεψη με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα δημιουργηθεί η απαραίτητη ε, εμπιστοσύνη ώστε να προχωρήσουν συμφωνίες όπως αυτές της, ε, των συμφωνιών START οι οποίες τελικά δεν ευδοκίμησαν. Δύο λεπτά απάντηση από την Επίτροπο την κυρία Άστον. Σας ευχαριστώ. Εγώ αγαπώ όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητος ο ενθουσιασμός που έχετε και θα επιτύχουμε έτσι τον ποινικό αφοπλισμό. Αυτό ήθελα να σας πω. Είναι απαραίτητο λοιπόν να έχουμε τον ενθουσιασμό να κινηθούμε προς την κατεύθυνση <clears throat> αυτή. Μπορεί να μην συμφωνούμε για το πώς θα γίνει κάτι τέτοιο, αλλά συμφωνούμε για το στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε. Και νομίζω ότι οι δηλώσει του Πρόεδρου των ΗΠΑ έχουν σημασία. Τώρα δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε εμεί να αντιμετωπίσουμε την συνδιάσκεψη τη επαλήθευση, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τύχει συζήτηση με τα κράτη-μέλη και να δούμε αν μπορούμε να έχουμε μια ενιαία και σαφή θέση για τα ζητήματα αυτά. Είναι σημαντική όμως η συνδιάσκεψη και έχετε δίκιο που το θέτετε επιτάπητος. Καταρχήν υπάρχει ευρεία υποστήριξη στο να αντιμετωπιστεί με καλύτερο τρόπο αυτή η εφαρμογή της συμφωνίας με πολυμερή τρόπο. Δεν πρόκειται να πω ότι απέτυχε η Κοπενχάγη, αντίθετα από πολλούς από εσά, νομίζω ότι υπήρξαν πολλά θετικά πράγματα τα οποία προήλθαν από την Κοπενχάγη και είναι ένα πρώτο εφαλτήριο αλλά θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια για το τι θέλουμε, αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα πολυμερέ πλαίσιο για την επαλήθευση τη μη διασπορά. Είναι πολύ δύσκολο όταν έχουμε πολλέ εμπλεκόμενε πλευρέ και είναι απαραίτητο να ξέρουμε εκ των προτέρων ότι μπορεί να υπάρξει μια κοινή στάση. Θα πρέπει να βελτιώνουμε λοιπόν όλο και περισσότερο τη συνεργασία μα. Κάτι το οποίο εγώ θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι για όλες τις συνδιασκέψεις χρειάζεται μια καλή προπαρασκευή. Αυτό όμως το οποίο με ενθαρρύνει είναι και η πρόοδος για τη μείωση των οπλοστασίων, αλλά κυρίως και η στρατηγική ενατένιση για αυτήν την μείωση των οπλοστασίων. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι το τι γίνεται σε ορισμένα κράτη στον κόσμο και οι δυσκολίες δεν είναι μονάχα η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί πυρηνική ενέργεια πολιτικού χαρακτήρα για παραγωγή πυρηνικών όπλων, αλλά και άλλα συναφή θέματα τα οποία πρέπει να απασχολήσουν την ε, διάσκεψη για την επαλήθευση. Κόουαν, ένα λεπτό. Κυρία Αντιπρόεδρε, είπατε προηγουμένως Αναφερθήκατε λοιπόν σε θέματα τα οποία έχουν σχέση με την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύετε ότι έχουν υπάρξει νέα στοιχεία από πλευράς της, Ρωσική, της Ρωσίας ε, για νέες ε, θέσεις της χώρας αυτής σχετικά με την Λευκορωσία, την Ουκρανία και τις χώρες που ανήκουν στην λεγόμενη ε, γειτονία. Και θα ήθελα να μάθω αν οι πρόεδροι των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών με τη Ρωσία και την Ουκρανία μπορούν να υπολογίζουν στις υπηρεσίες σας και να μας προσκαλέσετε στη συνάντηση κορυφής, στις συναντήσεις κορυφής οι οποίες θα διεξαχθούν στο μέλλον. Δύο λεπτά θα απαντήσει η ε, υποψηφία. Κοιτάξτε, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορώ να δώσω μια συγκεκριμένη απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, σχετικά με τον αγωγό Nord Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Θα εξετάσουμε όλους τους αγωγούς. Δεν έχω ένα χάρτη μπροστά μου για να σας μιλήσω πληρέστερα. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε την ενέργεια και την προέλευση της ανέργειας για να καλύψουμε τις ανάγκες μας στο μέλλον. Ένα από τα κρίσιμα θέματα ασφαλείας είναι η ενέργεια φυσικά και το Κοινοβούλιο θα έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Είπα επίσης ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει σαν ένωση και αυτό έχει, δεν είναι αστείο. Από κοινού θα πρέπει εμείς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την προμήθεια ενέργειας για την Ένωση. Αυτή είναι η βασική αντίληψη την οποία έχω για το συγκεκριμένο θέμα και αυτό φυσικά επηρεάζει τις στρατηγικές σχέσεις που έχουμε με χώρες όπως η Ρωσία στο μέλλον. Για την Ουκρανία έχω ήδη αναφερθεί στη συγκεκριμένη χώρα. Πολλά θα εξαρτηθούν από το ποιος θα κερδίσει τις εκλογές και ελπίζουμε η Ουκρανία να μπορέσει να καλύψει τις οικονομικές της υποχρεώσεις στον τομέα της ενέργειας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσπαθεί να τους βοηθήσει. Θα δούμε ακριβώς πώς θα προχωρήσει η σχέση αυτή στο μέλλον. Για τη Γεωργία η επόμενη συνάντηση θα γίνει στη Γενέβη στις 28 του μηνός θα είναι εκεί ο αντιπρόσωπος, ο ειδικό του Προέδρου της χώρας, του Πρωθυπουργού μάλλον της χώρας. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο που παίζουμε στη χώρα αυτή ε, στα πλαίσια της παρακολούθησης ε, της μεθοριακής γραμμής και ε, στα πλαίσια του διαλόγου τον οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε εμείς ανάμεσα στους εμπλεκομένους. Περιμένουμε λοιπόν το τι θα γίνει στην Γενέβη και αυτό έχει άμεση σχέση και ε, με το τι θα γίνει με τη Ρωσία αργότερα. Λούνατσεκ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, <clears throat> κυρία Άστον. Έχετε στο παρελθόν υποστηρίξει πράγματα τα οποία για μας είναι πάρα πολύ σημαντικούς, σημαντικά σε εμάς ως πρασίνους. Παραγματικά χάρη το ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντικότερα από τις οικονομικές σχέσεις. Θέλω να τονίσω ότι από τη δική μου ομάδα όμως υπάρχει μια κάποια απογοήτευση για το γεγονός ότι εσείς δεν, δεν μπορείτε να μας παρουσιάσετε πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τα οράματά σας, για το ποια είναι ποιοι είναι οι στόχοι σας και το κριτήριο που θα ακολουθήσετε για την περίοδο αυτή που θα έχετε τον ρόλο του Υπουργού Εξωτερικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε μια ηγεσία από την πλευρά σας, μια ηγετική στάση, όχι μόνο να είστε ο εκπρόσωπος 27 κρατών. Θέλουμε να είσαστε μια δεσμευμένη γυναίκα η οποία αναγωνίζεται για την πολιτική ειρήνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την πρόληψη και την αποτροπή των συγκρούσεων. Με ποιο τρόπο θα το εξασφαλίσετε αυτό στα επόμενα πέντε χρόνια, Πού είναι οι απόψεις σας, τα κριτήριά σας, οι στόχοι. Αυτό δεν το έχω ακόμα αντιληφθεί. <clears throat> δύο λεπτά από την κυρία Άστον. Εντάξει, σε δύο λεπτά. Ήλπιζα θα μπορούσα να τα εξηγήσω αυτά στην Από αυτά που είπα στην αρχή. Να σας πω τι σκοπεύω για την εξωτερική υπηρεσία, να καταλάβετε τι εννοώ. Κυρίως εννοώ θέματα ασφαλείας με μικρό α. Γιατί εμείς ως Ευρώπη πρέπει να συνεννοηθούμε με τρίτες χώρες για την ενίσχυση της ασφαλείας και ως προς κλιματολογικέ κλιματολογικές αλλαγές και οικονομική ασφάλεια, πράγμα που σημαίνει επίσης και συνεργασία με τον Επίτροπο Εμπορίου και άλλους. Είναι θέμα αναπτυξιακό ασφάλεια που επιτρέπει στις χώρες μέλη βιώσιμη ασφάλεια, μόρφωση για τα παιδιά τους κλπ. Είναι θέμα επίσης του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε. Ώστε όταν κάποιος μπαίνει σε κάποια ευρωπαϊκή πρεσβεία, αντιπροσωπεία κλπ. να βλέπει ότι η Ευρώπη συλλογικά εκπροσωπεί εκεί τις αξίες αυτές και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα σταθερότερο κόσμο και αποτροπή συγκρούσεων λοιπόν και άλλα θέματα ασφαλείας όπως αντιτρομοκρατικά, ναρκωτικά κλπ. Και όλα αυτά σε συνεργασία με τους στρατηγικούς μας εταίρους που καμιά φορά θα συνεισφέρουν περισσότερο πολιτικά, άλλες οικονομικά και μερικές φορές και στρατιωτικά, αλλά σε συνεργασία ώστε να φανεί ότι υποστηρίζουμε μια καλύτερη ζωή για τους πληθυσμούς των χωρών στις οποίες παρεμβαίνουμε. Δύο λεπτά και πέντε δευτερόλεπτα βλέπετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βρισκόμαστε στο τέλος της ακρόασης αυτής. Τον ε, Δεκέμβριο στην ακρόασή σας μας φανήκατε ιδιαίτερα να έχετε μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ένα πράγμα μονάχα μου δημιούργησε εντυπώσεις είναι ότι εσείς θέλετε περισσότερα πράγματα ως ε, Υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ό,τι προηγουμένως φαινόταν. Θέλουμε να ξέρουμε από τη δική μας πλευρά ότι εσείς θα είσαστε στο εκπρόσωπο της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι θα λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή λέτε ότι θα συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο, αλλά δεν υπάρχει στην ομάδα σύνδεσης με την οποία εργαζόσαστε ούτε ένας κοινοβουλευτικός σε σχέση με αυτήν την ε, εξωτερική υπηρεσία. Εσείς είσαστε το πρώτο άτομο που έχει αυτό το αξίωμα, επομένως θα είναι καθοριστικός ο ρόλος σας και η στάση σας γιατί θα δημιουργήσει προηγούμενο για το θέμα αυτό. Επομένως θα πρέπει να είστε πραγματικά ιδιαίτερα φιλόδοξοι στα θεσμικά επίπεδα. Και μιλάτε στις ε, γραπτές σας απαντήσεις για το γεγονός ότι υπάρχουν δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Γίνεται κάτι τέτοιο. Εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν είχα μια τέτοια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική στο Αφγανιστάν. Αλλά είναι αλήθεια. Δύο λεπτά να απαντήσει η κυρία Άστον. Προσπαθώ να απαντήσω τα ερωτήματα σε ό,τι αφορά την ε, πολιτική γειτονία και την εξωτερική υπηρεσία. Δεν είναι ότι αυτά τα θέματα έχουν μετακινηθεί από μένα, απλώς είναι τόσο σημαντικά που απαιτούν ένα πλήρης απασχόλησης επίτροπο, αλλά δεν είναι διαφορετικά τα θέματα αυτά. Εγώ νομίζω ότι είναι θετικό το ότι υπάρχει πια ένας επίτροπος ο οποίος ασχολείται ειδικά με τα θέματα αυτά για να μπορεί να είναι παρόν πολύ περισσότερο από ό,τι μπορώ να είμαι εγώ παρούσα και να αντιμετωπίζει όλες τις χώρες αυτής της περιοχής. Θα προτιμούσα το Κοινοβούλιο να μου δώσει ένα κατάλογο προτεραιοτήτων που να αφήνει έξω κάποιες χώρες. Γιατί αλλιώ όλε οι χώρε είναι πραγματικά σημαντικέ. Εγώ προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο φιλόδοξη, αλλά συγχρόνω και ρεαλιστική για το τι πράγματι μπορώ να επιτύχω. <clears throat> και γνωρίζω ότι έχετε προσδοκίες και από την Κομισιόν και από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό το να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα λειτουργήσει μια τελείως νέα υπηρεσία με την, μέσα στην οποία θα συνενωθούν όλες οι πολιτικές μας στον εξωτερικό χώρο και να μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλα τα τεκτενόμενα σε καθημερινό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παίξουμε ένα, ειδικά, ένα ιδιαίτερα ενεργό ρόλο. Χρειάζομαι λοιπόν όσο δυνατόν περισσότερη συνεργασία και αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε η Κομισιόν να λειτουργεί μαζί με εμένα και τα 27 κρατη και τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τότε η άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνεται πολύ πιο ακουστή σε όλο τον κόσμο. Η Διευθυντήρια Επιτροπή δεν είναι τα άτομα τα οποία, κύριε Λάμστροφ, που παίρνουν πολιτικές αποφάσεις. Είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τις αλλαγές σε επίπεδο χρηματοοικονομικό και επίπεδο κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης που του προσωπικού της υπηρεσίας εξωτερικών υποθέσεων δεν είναι αυτοί που παίρνουν στρατηγικές αποφάσεις. Εγώ θα επανέλθω ενώπιον του Κοινοβουλίου πριν από τις τελικές αποφάσεις και νομίζω ότι έχω εξηγήσει τη στάση μου για τους επικεφαλής των αντιπροσωπιών. Εγώ γνωρίζω ότι ορισμένε φορές πρέπει να κινηθούμε σε διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά αναγνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σεβερίν, ένα λεπτό. Ε, Κυρία Άστον, παρακολούθησα αυτά τα οποία είπατε, όχι για να ελέγξω τις γνώσεις σας, αλλά για να μπορέσω να κατανοήσω σε ποια βάση και προς ποια κατεύθυνση θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε στο μέλλον. Θα συμφωνήσετε μαζί μου λέγοντας ότι οι εξωτερικές μας σχέσεις δεν θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις αλλά να αυτενεργούν εκ των προτέρων και απαιτείται όραμα για να το πετύχουμε αυτό και ξεκάθαρη στόχοι. Ξεκάθαρη στόχοι φυσικά σημαίνει κοινέ αξίες και αντίληψη της γεωπολιτικής μας ταυτότητας. Εφόσον συμφωνούμε με αυτά θα μπορέσετε να μας βοηθήσετε για να διαμορφώσουμε το όραμα αυτό πριν βελτιώσουμε την πολιτική μας στις εξωτερικές σχέσεις. Δύο λεπτά για να απαντήσει η Αντιπρόεδρος. Υποψηφία Αντιπρόεδρος. Ναι. Να, ένα ναι το οποίο πολλοί από εμά θέλαμε να ακούσουμε. Να πω ότι μερικές φορές η φύση της διατύπωσης των ερωτήσεων δεν μπορεί να μου δώσει τη δυνατότητα να απαντήσω με ένα ναι και ένα όχι. Είσαστε πολιτικοί άνδρες και γυναίκες και ξέρω ότι κάποιες από τις ερωτήσεις σας ε, ε, με οδηγούν στο να προσπαθήσω να απαντήσω με μία παράφραση. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ σημασία η σχέση μου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα συμφωνήσουν και οι πρόεδροι της Επιτροπής ε, Εξωτερικού Εμπορίου ότι Όλα αυτά τα οποία άκουσα σήμερα θα πρέπει να προσπαθήσω να τα συνδυάσω. Ξέρω ότι κάποιος από εσά σας απογοήτευσα, λίγο ή πολύ. Αυτό ναι. συμβαίνει και αυτό θα συμβαίνει κιόλα, γιατί όσο προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια κοινή αντίληψη για τα πράγματα, κάποιοι δεν θα είναι απόλυτα ικανοποιημένοι. Υπάρχει όμως εμπειρογνωμοσύνη σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αίθουσα αυτή, υπάρχει πολιτική βούληση και φυσικά είσαστε δημοκρατικά εκλεγμένοι, κάτι το οποίο δεν είμαι εγώ και γι' αυτό έχω ανάγκη από εσά. Και αυτό έχει, τη σχέση αυτή έχει ανάγκη και η κοινωνία των πολιτών στην Ευρώπη. Πρέντα ένα λεπτό. Στο Πρόεδρε. επίτροπεξ Επίτροπε, της ομάδας του ΕΛΚ, μετά από διαβούλευση των υπολείπων, μπορούμε να σας πούμε ότι εκτιμούμε ιδιαίτερο την παρουσία σας σήμερα, περισσότερο από εκείνη του Δεκεμβρίου. Καταρχάς, εκτιμούμε το ανοιχτό σας πνεύμα ως προς το δημοσιονομικό έλεγχο και την απαλλαγή. Και θα θέλαμε να σας ξανακούσουμε από αυτού με περισσότερες λεπτομέρειες Αντίθετα, μας απογοητεύσατε κάπως ως προς τις ακροάσεις των υπευθύνων για την εκπροσώπηση. Γιατί εδώ είναι θέμα θεσμικής λογικής. Αφού θεωρείτε λογικό να σας ακροώμεθα εσάς, θα ακροαστούμε και αυτούς. Τέλος, ένα ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, για τη συνεργασία μας τις επόμενες εβδομάδες πώς ακριβώς θα συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην προπαρασκευή της οργάνωσης της λειτουργίας της εξωτερικής υπηρεσίας πριν από τη δημοσίευση μιας επίσημης πρότασης του Συμβουλίου. Με ποιον ακριβώς τρόπο Φτάνουμε στην κατάληξη της διαδικησίας και μέχρι τις 4 η κυρία Άστον έχει χρόνο να δώσει απαντήσεις στις τελευταίες ερωτήσεις και σχόλια του κυρίου Πρέντα και να κάνει τα τελικά της συμπεράσματα, να βγάλει τα τελικά της συμπεράσματα. Έχετε το λόγο κυρία Άστον. Ευχαριστώ κύριε Πρέντα, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εγώ φυσικά θα είμαι υπόλογος απέναντι στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα και με τη συνθήκη, είναι πάρα πολύ απλό. Θα δούμε αυτό πώς ε, θα εφαρμοστεί και τι αναμένεται από μένα να κάνω. Αυτό θα τα δείξει ο χρόνος. Πάντως ε, υπάρχει, αν κατάλαβα καλά, κυκλοφορεί μία πρόταση να έχουμε μία πρώτη συνάντηση τον Μάρτιο για να εξετάσουμε αυτές τις λεπτομέρειες και υπάρχει και ένα ερώτημα για το αν θα εμπλακούν και ε, τα εθνικά κοινοβούλια. Εγώ ε, εξαρτώμαι από εσά. Το Συμβούλιο θα πάρει αποφάσεις για τα θέματα αυτά τον μήνα Απρίλιο, δεν έχει πάρα... δηλαδή σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια δυνατότητα και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια ημερομηνία συζήτησης ε, σημαντική για όλους. Εάν επιθυμείτε, κυρία Άστον, να κάνετε ένα γενικό σχόλιο για το σύνολο της ακροάσεως. Έχετε το λόγο, κυρία Άστον. Εδώ είμαι. Θέλω να κάνω μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έθεσαν ερωτήματα και πραγματικά το εννοώ όλους αυτούς που έθεσαν ερωτήματα γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτή η ακρόαση να είναι μια ακρόαση που έχετε δυνατότητα να μου θέσετε όλα τα ερωτήματα. Μπορεί να μην πήρατε τις απαντήσεις που θέλατε, αλλά αυτές είναι οι απαντήσεις που μπορούσα να σας δώσω σε αυτή τη χρονική στιγμή. Δεύτερον, θέλω να τονίσω και πάλι την προσήλωσή μου προς τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι έχει γίνει σαφές και από την θητεία μου ως Επιτρόπου. Εγώ θεωρώ ότι είμαι υπόλογο προ το Κοινοβούλιο και θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι ώστε να δυνατόν πιο συχνά ενώπιον του Κοινοβουλίου μέσα στα ανθρωπίνω δυνατά χρονικά όρια. Τρίτον, η συνεργατική αυτή διάθεση του πρόεδρου της Επιτροπής μεταξύ των ε, Επιτρόπων είναι κάτι που πρέπει να το δείτε με το σωστό τρόπο. Είναι μια προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ όλων μας και θέλω να εξασφαλίσω τη συνεργασία με όλους τους Επιτρόπους. Τέταρτον, αναγνωρίζω τη σημασία και την αξία του έργου του Συμβουλίου και την μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη και πείρα των ε, Υπουργών Εξωτερικών των 27 κρατών μελών. Θα συνεργαστώ μαζί τους για να μπορέσω να ευνοηθώ από την υποστήριξή τους και να μπορέσω να αντιπροσωπεύω αποτελεσματικά το έργο όλων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τελευταίο, όσο παράξενο και να σας φαίνεται, προσβλέπω στην επόμενη συζήτησή μας. Όσο περισσότερο αναπτύσσεται ο διάλογος μεταξύ μας, τόσο περισσότερο καταλαβαίνω τι περιμένετε από μένα και τόσο καταλαβαίνω ποια είναι τα θέματα τα οποία έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για σας. Αλλά ενδιάμεσα θα πρέπει να θεωρείτε ότι έχετε τη δυνατότητα να έρθετε να με συναντήσετε, να μιλήσετε μαζί μου για θέματα τα οποία σας ενδιαφέρουν, είτε σε προσωπικό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικών ομάδων και ελπίζω θα βρίσκεται πάντα ανοιχτή την πόρτα, μου ανοιχτή. Και θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε παρά τη σημαντική κακοκαιρία σήμερα. Σας ευχαριστώ και πάλι ήταν μια σημαντική χρονική στιγμή για μένα και πιστεύω ότι και για σας θα ήταν πολύ σημαντική και χρήσιμη.